Dear colleagues. Τι συνάδελφοι, Λαμπέρ. Θα ήθελα να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Ξέρω ότι θα συνεχίσετε να έρχεστε τα επόμενα λεπτά, αλλά ξέρω ότι ο Επίτροπος μπορεί να μας διαθέσει μόνο το χρόνο που, του έχω, που έχουμε προβλέψει και θέλω να του πω ότι είμαστε ευγνώμονες που μπόρεσε να έρθει διότι είμαστε στις συζητήσεις τώρα και τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο σκέλος της πολιτική συνοχής και έχουμε αποφασίσει όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και εμείς να θέσουμε διάφορα θέματα σχετικά με τις κλιματολογικές αλλαγές και καλό θα ήταν εάν μπορείτε να μας πείτε πώς εσείς βλέπετε αυτό το θέμα, πώς μπορεί να γίνει ε, πιο αποτελεσματικό και όχι μόνο να προστατεύσουμε ε, την Ευρώπη αλλά και να χρησιμοποιήσουμε όλες τις ε, ε, δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και να δούμε τις ευκαιρίες, τις προοπτικές. Είμαστε διαθέσιμοι για περαιτέρω συζητήσεις και <clears throat> θα θέλαμε να μας πείτε ακριβώς ε, τι είναι οι ε, άποψή σας για την ε, επόμενη πτυχή της εξελίξεως της πολιτικής αυτής και έτσι ζητώ στην Επίτροπο να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαι μαζί σας σήμερα εδώ και πρέπει να σας πω ότι ε, εάν μπορούμε να έχουμε ένα διάλογο, εγώ και οι υπηρεσίες μου είμαστε στη διάθεσή σας για να οργανωθεί ο διάλογος αυτός. Εάν κοιτάξουμε τη γενικότερη εικόνα, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινούσε ε, το τη συζήτηση του πολιετούς πλαισίου το ερώτημα για μένα ήταν πώς είναι ο καλύτερος τρόπος να δαπανίσουμε ε, τους πόρους των ε, ε, φορολογουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό και να αντιληφθούν οι ενδιαφερόμενοι ότι αξίζει τον κόπο να χρηματοδοτούν τις Βρυξέλλες για να υπάρξει στη συνέχεια χρηματοδότηση κάποιου τομέα. Και στο κλίμα αυτό της λιτότητος είναι πολύ βασικό να εξετάσουμε τις πτυχές οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνες από τις χώρες και θα, γίνουν, θα είναι πιο αποτελεσματικά αν το κάνουμε μαζί. Δηλαδή, που θα υπάρχει μία σαφής ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Κάτι άλλο είναι οι δραστηριότητες ε, τις οποίες μπορούμε να εντείνουμε σαν πολιτικούς στόχους. Όταν δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση πρέπει να είμαστε ε, έξυπνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ε, ε, ξοδεύουμε κάτι για έναν στόχο αν μπορούμε συγχρόνως ε, να συγχρηματοδοτήσουμε και άλλους στόχους. Εάν δηλαδή βοηθούμε και τη γεωργία μέσω μιας υποδομής, μέσω ενός κτηρίου, θα ήταν σκόπιμο από την αρχή, από τη διάθεση των πόρων να προβλέψουμε ότι ήδη έχουμε κοιτάξει ένα πρόγραμμα και ε, προβλέπεται κάτι για τα επόμενα έτη. Το ίδιο είναι και το μήνυμα που θα αναφέρεται στην ε, βραχυπρόθεσμη απασχόληση αλλά που θα έχει και μακροπρόθεσμους στόχους διότι πιστεύω ότι θα πρέπει στην ευρωπαϊκή πολιτική να λάβουμε υπόψη και να συνυπολογίσουμε όλα αυτά τα θέματα κατά τρόπον ώστε να υπάρχει μία συνεκτική αντιμετώπιση και η δράση στον τομέα του κλίματος ε, ε, προσφέρει μία ε, αηφόρα κινητικότητα, βιώσιμες μεταφορές, υψηλότερη ενεργειακή ασφάλεια και θα οδηγήσει σε μικρότερη εισαγωγή ενεργειών και περισσότερα ωφέλη, καθαρότερο νερό, αέρα κτλ. Εάν ε, δε όλα αυτά γίνουν έξυπνα θα αυξηθεί και η ανταγωνιστικότητά μας. Γι' αυτό και ε, ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες για τις μελλοντικές εξαγωγές διότι ήδη χρησιμοποιούμε 3,5 ε, εκατομμύρια Ευρωπαίους στους οποίους απασχολούμε σε αυτούς τους τομείς και υπάρχει ενέργεια για τις οικογένειες, για τις επιχειρήσεις η ε, λογαριασμοί μας αυξάνονται και πρώτη φορά ε, φέτος ε, η μέση τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 ευρώ πράγμα το οποίο οδήγησε σε αντιδράσεις στην Ευρώπη διότι η τιμή που πληρώνουμε για το πετρέλαιο και μόνο αυξήθηκε 40% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ε, πρόπερς είχαμε δαπανίσει 315 δισεκατομμύρια στις εισαγωγές πετρελαίου. Ενδέχεται να σας φέρετε πολύ ψηλό το ποσό, αλλά ε, ποιος ξέρει πόσα είναι τα 315 δισεκατομμύρια, σχεδόν το ελληνικό ο χρέος, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός και βλέπουμε ότι ε, το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής ε, Ενώσεως ε, πέρυσι ήταν πάνω από ένα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή η εισαγωγή πετρελαίου κάλυψε όλα τα ωφέλη των ε, εξαγωγών μας προς άλλες χώρες. Άρα πρέπει να βελτιώσουμε τις μακροοικονομικές συνθήκες στην Ευρώπη. Ε, πρέπει επίσης ε, να υπάρξει ε, μία πρόθεση με τον τομέα ο οποίος είναι πολύ σημαντικός κατά τρόπον ώστε να διατηρήσουμε δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας και να έχουμε εξοικονόμηση τουλάχιστον 100 ευρώ ανά νοικοκυριό στην Ευρώπη. Αλλά ε, όλα αυτά δεν είναι τζάμπα. Χρειάζεται να υπάρξουν σημαντικές επενδύσεις που θα διατεθούν τα επόμενα έτη και αυτό θα πρέπει να καλυφθεί ιδίω από τους ιδιώτες επενδυτές αλλά και ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δαπανηθεί στις περιφέρειες όπου μπορεί κανείς να προκαλέσει αλλαγές γιατί τώρα 5% του προπολογισμού έχει σχέση με το κλίμα αλλά είναι πολύ περιορισμένος για να προκαλέσει διαρθρωτικές αλλαγές στις οικονομίες. Γι' αυτό και προτείνουμε να αυξήσουμε τις δαπάνες αυτές τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων. Δηλαδή, ε, θέλω να είμαι σαφής. Δεν σημαίνει ότι το ποσό αυτό θα, ασχοληθεί, θα αφιερωθεί μόνο στο κλίμα αλλά σε θέματα της ε, ε, της βελτιώσεως των κτηρίων για να αντέχουν στις κλιματολογικές αλλαγές ή σε βελτίωση των μεταφορών, των δημοσίων μεταφορών σιδηροδρομικών ή άλλων και επίσης να στηρίξουμε μία μετακίνηση προς μία οικονομία η οποία θα αντέχει στις κλιματολογικές αλλαγές και θα μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Μπορούμε να αναπτύξουμε καθαρότερες μεταφορές, να βελτιώσουμε ε, τα δίκτυα να είναι καλύτερα, να ε, διερευνήσουμε ε, πράσινες τεχνολογίες, να δημιουργήσουμε παράσινες θέσεις εργασίας, να έχουμε μία αναβάθμιση των δεξιοτήτων και όλα αυτά μπορούν να γίνουν αποκεντρωμένα. Συγχρόνως πρέπει να βελτιώσουμε τις ευρωπαϊκές στρατηγικές ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρειαστεί όλες τις δυνατότητες. Χρειαζόμαστε μία θεματική συγκέντρωση, μία ευξημένη ευελιξία για την περιφέρεια και πιστεύουμε ότι όλα αυτά αποτελούν μια καλή βάση. Ε, τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας ε, για να βελτιώσουμε τη τα κοινά ωφέλη. Καταρχήν πρέπει να επιτύχουμε ε, καλά αποτελέσματα στην πολιτική συνοχή με την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων με τις περιφέρειες και τα κράτη κατά τρόπον ώστε να επηρεάσουμε ε, τις επιπτώσεις της ευρωπαϊκής επέμβασης και αυτό θα, θα επιτευχθεί με την ε, νέα στρατηγική μας όπως αυτή της βιώσιμης ανάπτυξης. Πώς όμως ε, θα αυξήσουμε επενδύσεις οι οποίες είναι εκτός ε, αυτού του πλαισίου αλλά θα προωθήσουν ε, την πράσινη ανάπτυξη. Θα χρειαστούν όπως είπα περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις αλλά η πολιτική συνοχή δεν είναι ο μόνος τρόπος για τη χρηματοδότηση της Ευρώπης είναι λογικό και ιδίω ε, για αυτούς που πληρώνουν ε, τις πολιτικές αυτές να ε, χρησιμοποιηθεί χρηματοδότηση τους χώρους που εποφελούνται καλύτερα από αυτή τη χρηματοδότηση. Και ελπίζουμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα διότι υπάρχουν πολλά τα οποία προωθούν τις δικές τους πολιτικές ε, λόγω προσωπικών σκοπιμοτήτων, επερχομένων ε, εκλογών κτλ. Ενώ εμείς πιστεύουμε ότι εάν υπάρχει ένας καλός διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Περιφερειών θα επιτύχουμε πολλά περισσότερα. Για να μετρήσουμε τις επιδόσεις χρειαζόμαστε στόχους ε, σχετικά με τα αποτελέσματα των πολιτικών διότι στο τέλος η Επιτροπή και οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να ξέρουν μόνο τι ποσό δαπανήθηκε αλλά τι ε, επετεύχθη με αυτή την προσπάθεια δηλαδή βελτίωση του κλίματος, μείωση ε, της ρηπάνσεως και έτσι θα προσελκύσουμε στο μέλλον ε, περισσότερους που θα επενδύσουν στους στόχους μας και έχουμε πει ότι είμαστε καλύτεροι στις εφαρμογές. Δεν φτάνει κανείς να κάνει μεγαλοσχήμονες ε, δηλώσεις αλλά πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και ε, πώς επηρέασε την κατάσταση η χρηματοδότηση. Οι στόχοι θα επιτευχθούν εάν έχουν ε, καλυφθεί οι προϋποθέσεις. Θα πρέπει δηλαδή να ξέρουμε πώς θα υπάρχουν περισσότερα ωφέλη και θα γίνει μία ερεσιμότης εξ άντε κατά τρόπον ώστε να μπορέσουν τα κράτη να μεταφέρουν τις, στρατι τις οδηγίες ε, να τις εφαρμόσουν όσον αφορά την, την ανανέωση των ενεργειακών πηγών ε, και την βελτίωση του περιβάλλοντος ε, θα πρέπει να προσαρμοστούμε, να προσαρμόσουμε και τις ε, ε, τις ε, επενδύσεις μας ε, να έχουμε περισσότερες δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε τις θεομηνίες ε, και τις, τα πρόβλεπτα φαινόμενα. Θα πρέπει επίσης όταν προετοιμάζουμε και καταρτίζουμε προγράμματα να εξετάσουμε όλες τις πτυχές. Δεν θέλουμε δηλαδή να υπάρξει ένας σιδηρόδρομος που θα δια τρέχει μία ακτογραμμή η οποία ενδέχεται σε 20 χρόνια να έχει κατακλειστεί από τη θάλασσα. Πρέπει να βρούμε έξυπνους τρόπους να χρησιμοποιούμε τα χρήματα των φορολογουμένων. Θα πρέπει να προβούμε σε προσαρμογές που θα επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που έχουν σχέση με το κλίμα, να δούμε δηλαδή σε άλλες παρεμφερείς περιοχές πώς λύθηκε το πρόβλημα και πώς μπορούμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Τέλος, το πλαίσιο αυτό το οποίο ε, ε, επικεντρώνεται στους πόρους ε, θα ε, φροντίσει οι πόροι να διατεθούν σε στόχους που έχουν σχέση με την ε, στρατηγική του 2020, την καινοτομία, την έρευνα, τις επενδύσεις για χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, για προώθηση των νεοσύμων πηγών ενεργείας και θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι μία ροή και απαντούν στις ε, ανάγκες και πιστεύουμε ότι με το Ταμείο Συνοχής θα συμβάλλουμε στην κάλυψη των αναγκών κατά αυτόν τον τρόπο. Ε, θα μου πείτε δεν είμαστε πολύ άκαμπτοι. Όχι, καταρχήν τα επίπεδα είναι χαμηλά, άρα μπορούμε να τα πετύχουμε. Γι' αυτό και δεν πρέπει να, ε, ε, να υπάρξει διάχυση, διότι είτε πρόκειται για επένδυση στην υποδομή, στις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας ή σε οποιοδήποτε χώρο θα συνυπολογιστεί στο τελικό αποτέλεσμα για να επιτύχουμε τους ενεργειακούς στόχους και στους στόχους για την ε, ε, ε, ανανέωση για την ενέργεια για το περιβάλλον για το κλίμα τομείς που έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ λόγω της γραφειοκρατίας και χωρίς να έχουμε ένα τέτοιο σήμα για το μέλλον θα προσκρούσουμε στα ίδια προβλήματα και ε, ε, στο μέλλον αν δεν έχουν προσαρμοστεί οι αρχές εγκαίρως. Γι' αυτό <clears throat> και ε, θα σας πω ότι έλαβα μία επιστολή από την Συνέλευση Ευρωπαϊκών περιφερειών που στηρίζουν αυτό το σκεπτικό και τη δυνατότητα της ε, διοχετεύσεως των κλιματολογικών στόχων στον προϋπολογισμό ε, και ήταν μια στήριξη την οποία χαιρέτησα από αυτή την αρχή και ε, καταλήγοντας σας λέγω ότι ε, ε, ο, ίσως τα στοιχεία είναι πολύ λεπτομερή αλλά προσβλέπω στο διαλογό διότι πρέπει να προωθήσουμε έναν προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δείξουμε εις τους πολίτες ότι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις τις οποίες μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει να προσεγγίσει στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Έχουμε μισή ώρα αγαπητοί συνάδελφοι και θα ήθελα να κλείσω τον κατάλογο των αγοριτών έτσι ώστε να ξέρουμε ε, πόσοι θα είναι αυτοί που θα πάρουν τον λόγο. Επομένως, ε, ε, να δούμε πόσοι και ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να μιλήσουν. Θα ξεκινήσουμε τώρα με την κυρία Βέλτερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερος και την κυρία Χέντεγκαρτ που ήρθε σήμερα να μας ε, μιλήσει. Ε, ε, πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή της και την ευχαριστώ πολύ όπως την ευχαριστώ και για τη δουλειά της για τον Durban 2. Και πραγματικά παρακολουθούσαμε με μεγάλη ικανοποίηση την προσπάθειά σας. Ήδη ε, αναφερθήκατε και στο κόστος, το χρηματικό της κλιματικής αλλαγής. Ξέρουμε τι μας έχει κοστίσει και υπολογίζουμε και τι θα μας κοστίσει. Ε, υποψιάζομαι όμως ότι δεν έχετε συμπεριβάλει, συμπεριλάβει συγγνώμη, σε, αυτήν, σε αυτόν τον υπολογισμό ε, της, το κόστος της απώλειας της βιοπικιλότητας. Αυτή η απώλεια της βιοπικιλότητας έχει ήδη σημειωθεί ε, και όπως έχει πει και ένας άλλος συνάδελφος από όλη Επιτροπή είναι η σιωπηλή κρίση ε, Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία συνδυάζονται και σχετίζονται ε, με την απώλεια της βιοπικιλότητας και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βλέπουμε ας πούμε ότι λόγω της ε, ξηρασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Έχουμε ήδη απαγόρευση χρήσης ε, του νερού για συγκεκριμένες ώρες. Όλα αυτά έχουν προκληθεί από την κλιματική αλλαγή και βεβαίως αντίθετα και αντίστοιχα και το πρόβλημα των πλημμυρών. Υπάρχουν επίσης πολλά είδη ε, τα οποία θα ε, μετακινηθούν, ε, θα αποδημήσουν από την Ευρώπη και αυτό θα είναι μια μεγάλη απώλεια. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνυπολογιστεί στο οικονομικό κόστος. Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν έχετε συμπεριλάβει αυτού του είδους τα κόστη στους υπολογισμούς που κάνετε και επίσης με ποιο τρόπο μπορούμε να μετριάσουμε την κατάσταση, να προστατέψουμε την φύση, να κάνουμε πιο ε, αηφόρο την βιοπικιλότητα. Έχω 10 εγγεγραμμένους, λέει η Πρόεδρος, επομένως 1,5 λεπτό ο καθένας. Παρακαλώ πολύ να εστιάζετε στην ερώτηση που θέλετε να απευθύνετε προς την Επίτροπο, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα έστω για μία σύντομη απάντηση. Ε, κυρία Κρέλ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εσάς κυρία Επιτροπέ. Πολύ ενθουσιώδης η παρουσίασή σας. Ως συνεισηγήτρια για το γενικό κανονισμό θα ήθελα να κάνω την εξής παρατήρηση. Αν ήμουν στη θέση σας θα ήμουν και εγώ ευτυχής για την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής για την πολιτική συνοχή. Γιατί έτσι, σε, με μια πρόχειρη εκτίμηση πάνω κάτω τα λέει όλα για το κλίμα και τα χρηματοδοτεί. Εγώ δεν γνωρίζω κανέναν που να είναι κατά της προστασίας του κλίματος και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και των μέτρων. Αλλά εμείς εδώ είμαστε πολιτικοί, ε, άνδρες και γυναίκες αρμόδιοι για την πολιτική συνοχή και θέλω να το πω ξεκάθαρα. Η πολιτική συνοχή δεν ταυτίζεται με την προστασία του κλίματος. Βεβαίως πολλά μπορούν να συνδυαστούν και οφείλουν να συνδυαστούν έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά χρήματα, τα λεφτά των φορολογουμένων να πιάνουν τόπο. Αλλά ανάμεσα στην πολιτική συνοχή και την κλιματική αλλαγή και προστασία του κλίματος υπάρχουν και κάποιες διαφορές. Γι' αυτό μετά τις συζητήσεις που κάνουμε εδώ ε, στις επιτροπές, εβδομάδες ολόκληρες και μήνες, δεν το θεωρούμε ε, να αρκεί αυτό το θέμα της ευελιξίας της πιο ανεπτυγμένης περιφέρειας. Τα γνωρίζετε κι εσείς στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις νέες τεχνολογίες. Ε, υπάρχουν ορισμένοι που υπερβάλλουν. Παράδειγμα, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στην πόλη μου, έχουμε ένα εργοστάσιο βιομάζας παραγωγής ε, ενέργειας ηλεκτρικής, αλλά είναι ε, ε, πραγματικά ε, ικτρή κατάσταση οικονομικά γιατί χρησιμοποιεί πέλετς ξύλου που έχει εκτοξευτεί η τιμή τους στα ύψη. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι πάντα πιάνουν τόπο αυτά τα μέτρα και είναι τα σωστά. Η πολιτική συνοχή έχει να κάνει με μια συνοχή και δαυκή και κοινωνική και οικονομική και χάνεται καμιά φορά ε, σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και την καταπολέμησή της. Χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία ε, για τις περιφέρειες ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε περιφέρειας και θα πρέπει να μπορέσουμε με ευφύ τρόπο να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Κωνσταντίνε, σε αγαπώ πολύ, αλλά μίλησε πάνω από 2 λεπτά, 2 και 20 και ο Γιάννη Όμπριχτ να είναι κάτω από 1,5 λεπτό για να προλάβουμε. Uh, uh, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Επίτροπε για τα όσα μα είπατε και τον ωραίο τρόπο με τον οποίο τα παρουσιάσατε. Μια ερώτηση σχετικά με το RDF. Ποια είναι η άποψή σας ε, για το κείμενο που λέει ότι στις πιο αναπτυγμένες περιοχές ε, το ε, μέσω αυτό δεν θα στηρίξει περιβαλλοντικές υποδομές, υποδομές μεταφορών κτλ. Και ότι δεν θα αναπτυχθούν περαιτέρω όλες οι υποδομές οι οποίες αφορούν την μείωση του φαινομένου θερμοκηπίου κτλ. Ε, και επίσης την τέταρτη, ε, ε, στο τέταρτο συμπέρασμα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και της πολιτικής για περιβάλλον χωρίς διοξείδιο του άνθρακα ε, δεν καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ε, περί τίνος πρόκειται. Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν ε, θα πρέπει να πείτε ότι εάν μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι στο 80% δηλαδή των περιοχών δεν θα υπάρξει καθόλου επένδυση για προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και ότι θα απαγορευθούν η περαιτέρω, θα απαγορευτεί η περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών σε αυτές τις περιοχές, μα είναι το 80% 100%. Θα πρέπει να το ξαναδούμε, να είμαστε πιο ε, ευέλικτοι. Ευχαριστώ πολύ, ε, κυρία Επίτροπε ε, θα ήθελα και εγώ. Ευχαριστώ. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις κλιματολογικές αλλαγές, αλλά πρέπει να δούμε ότι ε, εδώ προσπαθούμε να μειώσουμε τις εκπομπές κατά λίγα ποσοστά, ενώ οι μεγάλοι ρηπαντές είναι εκτός Ευρώπης και δεν μας βοηθούν. Η πολιτική συνοχή μας βοηθάει για να μπορέσουμε να ε, εξισώσουμε τις ε, συνθήκες μεταξύ κρατών ε, αλλά υπάρχουν διαφορές μεταξύ των παλαιών κρατών μελών και των νεωτέρων και βλέπουμε ήδη το κόστος εργασίας και το κόστος ε, αποδόσεως το οποίο είναι πολύ ψηλότερο στην Ευρώπη από όπου αλλού. Γι' αυτό και φεύγουν οι επιχειρήσεις και παράγουν εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Άρα εσείς πώς διαβλέπετε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Διότι μιλάμε για τον ανταγωνισμό και εντό Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά και ακόμη περισσότερο για τον ανταγωνισμό μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ε, ε, μάλλον ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εις την διεθνή σκηνή γιατί πρέπει να σκεφτούμε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σχετικά με το τελευταίο ζήτημα, δηλαδή που βλέπω να υπάρχουν θέσεις εργασίας, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο λόγος για τον οποίο ε, ανέφερα αυτό το αριθμητικό στοιχείο για τις εισαγωγές ε, ε, πετρελαίου ε, μία άποψη βεβαίω καταδεικνύουν πόσο εξαρτημένοι είμαστε από τι εισαγωγέ. Όμω, εάν κάνουμε την οικονομία μα πιο αποτελεσματική από άποψη ενεργειακή, τότε οπωσδήποτε θα εξοικονομήσουμε χρήματα. Είναι επίση σαφέ ε, ότι ε, όταν προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις, ε, την τροφοδοσία των κτηρίων, τις σωληνώσεις και τα τότε οπωσδήποτε μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας οι οποίες δεν μπορούν μέσω εξωτερήκευσης του κόστους να αντικατασταθούν. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να υποκαταστήσει αυτή τη δουλειά δουλειά με κάτι που εισάγει από την Κίνα ή κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λοιπόν ε, είναι κάτι το οποίο εδώ τοπικά, περιφερειακά μπορεί ε, να δώσει όθηση στην δραστηριότητα και ταυτοχρόνως στην απασχόληση και ταυτοχρόνως να έχει και ένα μακροχρόνιο αντίκτυπο και να μας βοηθήσει να εξοικονομήσουμε χρήματα. Πιστεύω ότι με τον ίδιο τρόπο και την ίδια λογική ε, θα δώσει νέα όθηση και στην οικονομία ε, και την καινοτομία, συγγνώμη, γιατί χρειάζεται και νέα τεχνογνωσία έτσι ώστε ε, να αποκαταστήσει κανείς ε, συστήματα τροφοδοσίας και και επομένως μπορούμε να αυξήσουμε την καινοτομία και ταυτοχρόνως να αυξήσουμε την εξαγωγή τέτοιων καινοτομιών. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μόνο. Ε, κύριε Όλμπρεχτ, αναφέρθηκε στις μεταφορές και γιατί, ο, κύριος μάλλον, η, η, λογική της πρότασης Επιτροπής ε, ήταν ότι αναφερόμαστε ε, περισσότερο σε υποδομή που έχει να κάνει με τα κέντρα ε, της, της ενέργειας, grids λοιπά. Δεν μιλάμε πολύ για την ε, μεταφορά και ούτως ή άλλως ε, όταν μιλάμε για, το, για μεταφορά μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα ε, ποσά και τότε σε αυτή την περίπτωση ναι, ίσως να χρειαστούν και άλλα χρήματα γιατί ε, ε, τα, τα πρώτα χρήματα θα δαπανηθούν οπωσδήποτε ε, για προγράμματα ενεργειακής επάρκειας. Μην ξεχνάτε ότι οι στόχοι του 2020 δεν είναι καινούργοι. Ήδη από το 2008 είχαμε αποφασίσει ότι θα έχουμε το 10% της βελτίωσης και παρόλα αυτά φτάνουμε τώρα στο 8%. Ε, είπατε επίσης ότι δεν μπορεί να έχουμε πολιτική συνοχή σε η οποία να βασίζεται, η κυρία Κρέλ το είπε αυτό, η οποία να βασίζεται μονάχα ε, στην ε, κλιματική αλλαγή. Ναι, εντάξει, πρέπει να πω ότι είμαστε και πρέπει να έχουμε ευελιξία. Εγώ λέω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την ευελιξία. Έτσι το είδαμε τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορώ να καταλάβω βέβαια γιατί ορισμένα κράτη-μέλη ζητούν ευελιξία. Αυτή τη στιγμή συζητούμε είναι τον κανονισμό της ενεργειακής ασφάλειας ε, επάρκειας και όλοι λένε θα έχουμε ευελιξία. Ναι, αλλά τι σημαίνει αυτή η ευελιξία. Το, το θέμα είναι αν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας ή όχι και, και σε αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς ε, γιατί καμιά φορά πίσω από τον όρο ευελιξία κρύβεται η πρόταση θα κάνουμε τελικά ό,τι θέλουμε. Ε, επομένως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έχουμε ένα προπολογισμό, έχουμε μια δέσμευση και με τα κράτη-μέλη. Και επομένως ε, θα, θα δαπανηθούν ευρωπαϊκά χρήματα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο εάν είμαστε σίγουροι ότι θα επιτύχουμε ε, με τη δαπάνη των χρημάτων αυτών τον πολιτικό στόχο τον οποίο έχουμε ήδη θέσει. Είναι πολλές και διαφορετικές οι προτεραιότητες, ε, είναι διάσπαρτες στις διάφορες χώρες αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει κάθε φορά και σε κάθε περίπτωση να αποδεικνύουμε στον Ευρωπαίο πολίτη ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία, ότι αξίζει τον κόπο και επομένω έτσι να αποκτήσουν έννοια όλα αυτά τα πράγματα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Όσον αφορά τώρα το κόστος της ε, απώλειας της ε, βιοπικιλότητας και ε, σε σχέση με, την, με τον υπολογισμό του κόστους της κλιματικής αλλαγής. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να βρούμε και να συνυπολογίσουμε και κάποια επιπλέον ωφέλη από τον καθαρότερο αέρα κτλ. Όμως έχετε δίκιο που λέτε εδώ ότι η βιοπικιλότητα ε, έχει και οικονομικό ε, αντίκτυπο Ε, και θα πρέπει να συνυπολογιστούν τα κόστη. Αυτά που ε, αυτό που κάνουμε και στον εξωτερικό προϋπολογισμό και ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και εγώ προσπαθούμε να δούμε ε, την, το, την, τη διασύνδεση που θα μπορούσε να υπάρχει ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή και την βιοπικιλότητα. Σαν Ευρώπη δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που πάμε σε μια νέα ε, διεθνή διάσκεψη να ζητάμε νέα χρήματα, καινούργια χρήματα για την ενέργεια, καινούργια χρήματα για το ένα, καινούργια χρήματα για το άλλο. Και επίσης ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε με πιο ολιστικό τρόπο να δούμε τα πράγματα, δηλαδή να προτείνουμε κάτι το οποίο θα είναι καλό συνολικά. Ευχαριστώ πολύ. Λαμπερ Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε. Πολύ ορθά μιλάτε σε σχέση με την δέσμευση των ε, κρατών ε, μελών και, τους, ε, και των πολιτών στην σωστή ημερήσια διάταξη. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κατακαιρματισμός των δαπανών. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική, μια σφαιρική προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα και νομίζω ότι η προσέγγιση αυτή είναι ισχυρή. Ε, Υπάρχει εδώ όμως μια παγίδα, λέτε ότι ένα και ένα θα κάνουν τρία, αλλά υπάρχει και μια παγίδα και μπορεί το ένα και ένα τελικά να ε, ε, κάνει άθροισμα μηδέν, δηλαδή δίνουν διαρκώς περισσότερα χρήματα, αναγκαζόμενοι να κόψουν, ε, να κάνουν περικοπές από την έρευνα και την ανάπτυξη, από κάποια άλλα προγράμματα και παρότι λοιπόν συμμερίζομαι το πάθος σας και τη δουλειά σας στο Συμβούλιο, πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε ε, να ε, μην λάβουμε υπόψη μας το θέμα της ενεργειακής απόδοσης για τα κράτη και για τα νέα κράτη-μέλη. Και ε, το, το ζήτημα είναι όχι μόνο να βρούμε τα αριθμητικά στοιχεία, αλλά να δούμε πώς τι, θα τα κάνουμε τα αριθμητικά αυτά στοιχεία, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσετε τα οικονομικά κίνητρα. Στην Ελλάδα, ας πούμε υπάρχει μεγάλη ε, ανάγκη και μεγάλες ευκαιρίες ε, για επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ε, ιδίως δε στην ηλιακή ενέργεια. Ε, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα γιατί διαφορετικά πώς θα επιτύχετε τους στόχους σας Ευχαριστώ η κυρία Σμόκοβα Ευχαριστώ Πρόεδρε Σύντομα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, για ε, τα όσα μας είπατε, για ε, την πειθαρχία βεβαίως και για τη σωστή χρήση των πόρων. Έχω μια ερώτηση. Την περασμένη εβδομάδα συνεδρίασε στη Μασαλία το Παγκόσμιο Φόρουμ για το νερό. Και ξέρουμε ότι αυτό συνδέεται πάρα πολύ με την κλιματική αλλαγή. Ένα από τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής είναι η λειψιδρία. Αλλά αλλού κάθε χρόνο έχουμε πλημμύρες. Τι μέτρα συγκεκριμένα όμως έχετε καταρτήσει για να αντιμετωπίσετε αυτά τα φαινόμενα. Διότι πολύ συχνά ε, ο λόγος εδώ που αποτυχάνουμε είναι ακριβώς η έλλειψη πειθαρχία. Ευχαριστώ. Κυρία Σρότερ. Πολύ σύντομα. Πρώτον, θεωρώ σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν έκθεση για τις πράσινες λεγόμενες θέσεις εργασίας, green jobs και πολλά τα λέει η διέκθεσή μας από αυτά που είπε η κυρία Χέτεκα συμπεριλαμβανομένων και των διαρθρωτικών ταμείων που θα πρέπει ε, να έχουν συνδυαστική ε, δράση. Δηλαδή υπάρχει στο Κοινοβούλιο απόφαση σχετικά η ε, συγκεκριμένα για τον κανονισμό. Πρέπει να πω ότι το πρόβλημα είναι το εξής. Σε ορισμένες δομές του γενικού κανονισμού έχει γίνει κάποια παρεξήγηση και αυτή θα πρέπει να λυθεί αλλού, όχι στο 20%. Δηλαδή μπορούμε να φροντίσουμε περισσότερες πολιτικές, περισσότερη κλάδη πολιτικής να φτάσουν στο 20%. Και υπάρχει μια πρόταση να σκεφτούμε τι θα γίνει ε, με την αηφόρο ε, συγκοινωνία ή τις αηφόρες μεταφορές γιατί έτσι θα φτάσουμε ξέρετε ότι οι μεταφορές είναι μέγα τμήμα αυτού δηλαδή ανάμεσα στο 4 και στο 7 χρειάζεται μια αναδιατύπωση αν θέλετε και είναι πάρα πολύ σημαντικό το έχουμε συζητήσει και με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τότε πραγματικά θα φτάσουμε σε αυτό το στόχο γιατί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο Δεύτερον, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αν το κοιτάξετε, ακριβώς εκεί έχει εξαιρεθεί η ενέργεια και υπάρχει λόγος για την e, ε, το FES δίκτυο, το Smart Grid, χρειάζονται ειδικέ ε, ρυθμίσεις και επίσης ε, για θέματα του νερού. Υπάρχει και μια πρόταση της Επιτροπής Μεταφορών, την οποία θεωρώ πολύ καλή, εκεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης να φροντίσουμε να μπουν οι αϊφόρες αστικές συγκοινωνίες. Δηλαδή, να μπορεί να χρηματοδοτείται αυτή η προσπάθεια και να συνεισφέρει στο 20%. Αν τα συνδυάσουμε όλα αυτά και τα λύσουμε, τότε λύνουμε και το πρόβλημα και μπορούμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Ακριβώς αυτή είναι η ιδέα και ο στόχος, όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφικτός. Αυτά τα πράγματα δεν κολλάνε στο 20%. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, αλλά είναι ότι δεν έχουν μπει στη σωστή θέση του κανονισμού. Και επίσης η συγκέντρωση δεν θα πρέπει να είναι σε επίπεδο προτεραιότητας επενδύσεων, αλλά στους θεματικούς στόχους, για να έχουμε πολλαπλή χρηματοδότηση από πολλά ταμεία και να έχουμε και αυτό το στόχο και το αποτέλεσμα που πρότεινε η κυρία Χέντεγκαρτ. Και θα παρακαλούσα να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. είναι, δεν, είναι λιγότερο ερώτηση όλα αυτά που σας λέω, αλλά πρέπει να τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ, Βίκτορ Μποστινάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και κυρία Επίτροπε. Συγγνώμη που καθυστέρησα, γιατί στην Επιτροπή Αναφορών έχουμε, είχαμε μεγάλη ψηφοφορία. Θα ήθελα να σας... Σας ευχαριστώ ε, τώρα λοιπόν καλούμαστε να εγκρίνουμε κανόνες για το επόμενο διάστημα, την επόμενη προγραμματική περίοδο, ε, τις δημοσιονομικές και να βάλουμε και τη διάσταση του κλίματος. Είπατε προηγουμένως ότι είστε δεσμευμένοι, αλλά και τα κράτη-μέλη πρέπει να δεσμευθούν. Πέρυσι, σε μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώθηκε ότι με το σημερινό ρυθμό μπορούμε να φτάσουμε μόνο στα 10 σημεία στο 10% δηλαδή τη στρατηγική για το 2020 αντί να φτάσουμε στο 20%. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω τη δική μου δέσμευση να μπει στο Ταμείο Συνοχής ένα σύνολο προγραμμάτων και έργων που συνδέονται ε, με την εξοικονόμηση ενέργειας στη στέγαση, στα σπίτια και από την άλλη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας ε, στα εργοστάσια πάνω από 20 ΜΒ. Γιατί το λέω αυτό, έχω εδώ μια μελέτη. Δεν θα σας μιλήσω για τα ωφέλη από πλευράς κλιματικής αλλαγής και περιβαλλοντικής δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, μείωσης των αερίων θερμοκηπίου κτλ. Εκπομπές και πάει λέγοντας και εξοικονόμηση ε, χρημάτων από τους λογαριασμούς της ε, ενέργειας. Άλλο θέλω να σας πω. Γνωρίζετε την νέων ε, έχουν ένα κέντρο ερευνών για την ενέργεια και μετράνε το μέγεθος των μονάδων, των βιομηχανικών, όταν είναι μικρά τα εργοστάσια, είναι λιγότερη η αποδόση τους ε, σε σχέση με τα μεγαλύτερα εργοστάσια και γίνονται μεγάλες επενδύσεις. Ε, αν πηγαίνουν σε μικρές βιομηχανικές μονάδες είναι μεγαλύτερη η επιβάρυνση και ε, αυξάνεται το συνολικό συστημικό κόστος. Προτείνω λοιπόν το εξής ε, και θέλω και την υποστήριξή σας. Μπορούμε με κάποιο τρόπο να αλλάξουμε τους κανόνες για να επιτρέπονται και μεγαλύτερα εργοστάσια και εργοστάσια συνδυασμένη παραγωγής θερμότητας να είναι επιλέξιμα. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσουμε στους στόχους στρατηγικής του 2020. Αλλιώς θα έρθουμε και πάλι το 20 να ανακαλύπτουμε ότι αποτύχαμε. Αποτύχαμε, θα έχουμε αποτύχει, αλλά το κόστος θα επιβαρύνει τους Ευρωπαίους πολίτες. Όχι μόνο τα κράτη-μέλη, τους πολίτες πρώτα απ' όλα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι έτοιμος να ακούσω τα σχόλιά σας και όσο μπορώ να σας υποστηρίξω και εγώ από πλευράς μου. Ευχαριστώ πολύ. Η τελευταία ερώτηση ήταν αυτή, αλλά θα ήθελα να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, για την ανάγκη να έχουμε πολιτικές που να καταπολεμούν την κλιματική αλλαγή και να συνάδουν. Έχετε σκεφτεί δηλαδή να αναθεωρήσετε κάποιες οδηγίες ε, για τις μελέτες περιβαλλοντικού αντικτύπου, για την αξιολόγηση την περιβαλλοντική, γιατί έχουν και μια ιστορία αυτές οι οδηγίες πριν από την κλιματική αλλαγή υπήρχαν. Ε, για την τελευταία ερώτηση, Επίτροπος, το έχουμε σκεφτεί, αλλά είναι σαφές ότι και τα κράτη-μέλη όταν γνωρίζουν ας πούμε ότι θα αυξηθεί η στάθμη της θάλασσας, θα πρέπει να προγραμματίζουν λίγο περισσότερο συντονισμένα που θα χτίσουν. Όταν μπαίνει στο σχέδιο, ας πούμε, μια περιοχή, μιας πόλης δίπλα σε ένα λιμάνι, θα πρέπει ε, τα κτίρια να χτίζονται λίγο πιο ψηλά, γιατί θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας. Ε, του χρόνου θα έχουμε μια στρατηγική προσαρμογής και θα τα εντάξουμε ε, όλα αυτά στα ε, κείμενά μας και στις προτάσεις μας. Προσοχή όμως να μην είμαστε υπερβολικά περιοριστικοί στα όσα υπαγορεύουμε από το ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ε, στα κράτη-μέλη υπάρχουν μεγάλες διαφορές και ιδιαιτερότητες. Το 2013 αναμένεται το πρώτο τετράμινο ή το πρώτο τρίμηνο ε, μια τέτοια πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρου για τα σχόλιά σας. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε για τις μονάδες συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας υπάρχει δυνατότητα να μπει στο ΦΕΝΤΕΡ, ε, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά ξέρω ότι θέλετε να είναι και στο Ταμείο Συνοχής και τα θέματα των ε, εκπομπών ρήπου και της εμπορίας, τα είπε και η κυρία Κρέλ. Θα πρέπει να εστιάσουμε στο Ταμείο Συνοχής. Αυτό σας ενδιαφέρει σας. Καταλαβαίνω αυτά που λέτε, τα σημειώνω και θα τα ε, διαβεβάσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εσωτερικές ε, συζητήσεις που γίνονται. Η κυρία Σρότερ μίλησε για τις αηφόρες αστικές συγκοινωνίες και μεταφορές γενικά. Έχουμε στόχο στον προϋπολογισμό ε, αν θα πρέπει να είναι 20% παντού στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Στο ΕΤΠΑ είναι 6% και 20% αντίστοιχα. Εμείς εστιάζουμε σε αυτό που συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Ε, οι αηφόρες συγκοινωνίες δεν είναι ότι δεν λαμβάνονται υπόψη, αλλά δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες. Η κυρία Σμόλκοβα μίλησε για τις πλημμύρες, για τις πολιτικές υδάτων, ε, λειψιδρία κλπ. Ξέρω ότι ο Επίτροπος Ποτότσνικ, ο συνάδελφός μου του χρόνου, θα φέρει μια πρόταση για το νερό. Ακριβώς ε, πολλά από τα σημεία αυτά θα καλύπτονται εκεί και θα έχουμε και σχέδια ε, προσαρμογής. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να αλλάξουμε την εστίαση μας, τον τρόπο με τον οποίο ασχολούμαστε στην Ευρώπη με αυτά τα θέματα οι πολίτες θα ζουν όλο και περισσότερες πλημμύρες στην Ευρώπη, ενώ σε κάποια άλλα μέρη, στην Νότια Ευρώπη, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία, θα είναι πολύ περισσότερη λειψιδρία. Στην Πορτογαλία άκουσα ότι έχει να βρέξει από τον Νοέμβριο. Και ε, κανονικά η βροχοπτώση είναι το χειμώνα. Ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ορισμένες περιοχές τεχνικά περιγράφονται ως σε ξηρασία ήδη. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Η πρόταση για το νερό θα προσπαθήσει να λάβει υπόψη της αυτά τα στοιχεία της ανησυχίας, καλύτερη διαχείριση. Υπάρχουν ήδη πολιτικές που θα ε, προσπαθήσουμε να έχουμε πιο μεγάλη συνοχή σε αυτές. Τελευταίο για τον κύριο Βανίστερόι. Τι κάνουμε με το Συμβούλιο. Μας λέει τι νόημα έχει να έχετε ε, οικονομική συνεισφορά χωρίς τον κανονισμό. Μα γι' αυτό έχουμε και την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση. Πώς θα προτείνουμε τα έργα, τα μέσα, τα εργαλεία, τι χρειάζεται να γίνει, ποιες είναι οι προαπαιτήσεις. Θα πρέπει να πηγαίνουν χέρι με χέρι οι κανόνες με τον προπολογισμό. Αλλού είναι οι περιφερειακές αρχές που αποφασίζουν, αλλού οι τοπικές, αλλού οι εθνικές. Που μας λένε ότι είναι πάρα πολύ χαλεπή Μην μας ζητάτε να κάνουμε τόσα πράγματα. Πού θα βρούμε τα λεφτά. Έτσι θα πρέπει να συνδέουμε τις πολιτικές μας προτεραιότητες με τον προϋπολογισμό. Και ένα τελευταίο. Πιστεύω ότι είναι πραγματικά σημαντικό να προσπαθήσουμε και εσείς τελικά να προσελκύσουμε περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις. Βεβαίως δεν μπορούμε από το κρατικό προϋπολογισμό να ε, επισκευάσουμε και να ανακαινήσουμε όλα τα κτίρια θα πρέπει να προσελκύσουμε και ιδιωτικό κεφάλαιο. Μες δίτ, γιατί εκεί δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης. Τελειώνω, Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Σε ό,τι φορά τη συνέλευση των ευρωπαϊκών περιφερειών, μου έστειλαν μία επιστολή και λέγουν ότι μετά από τη διαβούλευση που είχαμε με τα μέλη μας, η Πρόεδρος ε, σας ενημερώνει ότι υποστηρίζουμε ε, αυτά τα ειδικά κονδύλια για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και χαιρόμαστε για την πρόταση των θεματικών στόχων στρατηγική του 2020 και αναγνωρίζουμε την επίγουσα ανάγκη να αντιδράσουμε, να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και ε, τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Το 20% του ΕΤΠΑ θα πρέπει να πηγαίνει σε μια οικονομία χαμηλής παραγωγής διοξιδίου του άνθρακα και θα μπορέσουν οι περιφέρειες να αναπτύξουν καινοτομία και βέλτιστες πρακτικές και ταυτόχρονα να εξοικονομούν εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα για μας που προσπαθούμε να βοηθήσουμε με αυτά τα προγράμματα. Ξέρω ότι καμιά φορά τα κράτη-μέλη θέλουν περισσότερη ευελιξία, και να αποφασίζουν εκείνα τι θα κάνουν οι περιφέρειέ του, αλλά οι περιφέρειες μα στέλνουν ένα πολύ σαφέ μήνυμα ότι υποστηρίζουν πολλές από τι δικέ μα πολιτικέ. Σα ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να έχω το διάλογο μαζί σα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ε, με συγχωρείτε. Ξέρετε όμως ότι έχετε πέραν των περιφερειών και άλλους σημαντικούς τομείς όπως είναι ε, οι πόλεις ε, όπου επίσης ε, η υπόθεση του κλίματος είναι σημαντική διότι στις πόλεις λέγεται ότι θα παιχθεί ή θα χαθεί η υπόθεση των κλιματολογικών αλλαγών. Ευχαριστώ.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 Όσον αφορά τις ε, κατηδίαν πρωτοβουλίες εκθέσεις, αποφασίσαμε να ζητήσουμε στις εκθέσεις κατά πρωτοβουλία την ε, ευρωπαϊκή πολιτική στα ε, πλαίσια της συνοχής θα αναλυφθεί από το ΕΛΚ και θα αποφασιστεί ο τίτλος οι κλιματολογικές αλλαγές και η δομή στο περιφερειακό επίπεδο όπως και η ακριβής διατύπωση θα αποφασιστεί αλλά σε αυτή, την, ε, αυτή θα είναι η δεύτερη έκθεση η τρίτη έκθεση είναι η έβδομη έκθεση προόδου και θα αναλυφθεί από τους φιλελεύθερους επίσης ε, ζητήθηκε να υπάρξει μία έκθεση για την εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ενώσεως, την οποία θα αναλάβει το ΕΛΚ μετά είπαμε για την κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Ήτρε για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης του 2020 στη διαρθρωτική ε, και περιφερειακή πολιτική και συμφωνήσαμε να γίνει ε, κοινά ε, από κοινού η ακρόαση αυτή στις 29 Μαΐου όταν ε, θα, ε, όπου θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 4.30 το απόγευμα. Πέραν αυτού, θα συνεχίσουμε για το δεύτερο ήμιση της ε, θητείας μας να εντοπιζόμαστε στην ισότητα των φίλων κατά τη διατύπωση των πολιτικών μας και συμφωνήσαμε ότι ε, η Ελίζα Σρότερ θα είναι η υπεύθυνη για την ε, εποπτεία η οποία ε, είχε παρακολουθήσει τον τομέα και κατά το, τα πρώτα δυόμιση χρόνια. Τώρα θα ψηφίσουμε. Καταρχής ελέξτε ότι έχετε τις κάρτες σας ψηφοφορίας και τα, ότι λειτουργούν σωστά τα μηχανήματά σας. Θα κάνουμε λοιπόν μια δοκιμαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία η οποία ξεκινά για έλεγχο. Ε, βλέπω ότι 40 έχουν βάλει τις κάρτες τους αλλά μόνο 36 ψήφισαν. Μπορείτε σας παρακαλώ να ψηφίσετε και οι υπόλοιποι. Ψήφισαν 37 ε, από τις 40 κάρτες της μηχανές. Ε, δεν ξέρω, οι άλλοι δεν ψήφισαν ή δεν λειτουργεί το μηχάνημά τους. Λειτουργεί. Οπότε ξεκινούμε τις ψηφοφορίες. Έχουμε ε, δύο έγγραφα το πρώτο είναι η συναπόφαση για τη συμμετοχή ή στην ανάληψη κινδύνων. Μπορούμε να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Οι διατάξει σχετικά με τα μέσα επιμερισμού κινδύνων και τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα. Ξεκινάμε λοιπόν με ε, τη συμβιβαστική 1. Ε, 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. στο άρθρο 2 υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Κάποιος έχει αντίρρηση, όχι, τότε την ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Νομίζω ότι δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Και με το φως που έχουμε εδώ και την αντιλιά δεν μπορούμε να δούμε. Προχωράμε στην τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. εκτιμώντας 3 προφορική τροπολογία κανείς δεν έχει αντίρρηση ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 1 ποιος είναι υπέρ της συμβιβαστικής 1 κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας 6 προφορική έχει κανείς ε, ε, αντίρρηση όχι τότε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψοφορική τροπολογία στο εκτιμώντας 11 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 22 Ποιος είναι υπέρ της ε, τροπολογίας 22. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, τροπολογία 6 με προφορική τροπολογία αν δεν έχει αντίρρηση την ψηφίζουμε ε, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην τροπολογία 8, ε, προφορική τροπολογία. Αν δεν έχετε αντίρρηση την ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9, προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τώρα πάμε στις ε, τροπολογίες Επιτροπής ε, Ελέγχου του Προϋπολογισμού. και ψηφίζουμε την τροπολογία 1 της Επιτροπής υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα πάμε στις ε, τροπολογίες για την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Ε, θα γίνουν ηλεκτρονικά οι ψηφοφορίες. Ψηφίζουμε, με συγχωρείτε, λάθος, προχωρούμε στην τελική ψηφοφορία ε, υπάρχει ένας ε, ΕΛΚ πλεονάζων και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την νομοθετική πρόταση όπως ε, τροποποιήθηκε εγκρίθηκε με 35 ε, υπέρ δύο, κατά και αποχές και ε, όσον αφορά το νομοθετικό ψήφισμα ψηφίσατε όλοι Δύο δεν ψηφίζουν, δεν ξέρουμε γιατί. Λίγοι. Τρεις δεν ψήφισαν. 36 υπέρ, 2 ε, κατά και 5 αποχές. Και εγκρίθηκε. Περνούμε τώρα στη δεύτερη ψηφοφορία. Ε, είναι η γνωμοδότηση του Νούνου Χέιρα ρόλο πολιτικής συνοχής στι ιδιαίτερα προγραμματισμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα πλαίσια της στρατηγική Ευρώπη 2020. Παρακαλώ. Θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η έκθεση αυτή. Δεν καταλαβαίνω γιατί ε, η συγγετρία, μάλλον ο εισηγητής δεν ε, ξεκίνησε νωρίτερα. Είναι, με ενοχλεί που την μετάφραση των πολλών τροπολογιών την είχαμε πάρα πολύ αργά την προηγούμενη Τετάρτη, ε, πράγμα που σημαίνει ότι δυσκολεύει πάρα πολύ την ε, την δουλειά μας ε, ε, και τα περισσότερα μέλη του Κοινοβουλίου έφυγαν την Τετάρτη του κοινοβουλίου χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν τις τροπολογίες αυτές. Δεν πρέπει με τον τρόπο αυτό να κάνουμε τις εκθέσεις. Δεν μπορεί να μην υπάρχει επίσης επίσημη μετάφραση για, τα, για τις συμβαστικές τροποποίησεις. Επίσης ε, δεν ε, υπάρχει καμία μετάφραση στα εστονικά. Ε, ούτε εδώ τώρα στην συνεδρίαση δεν έχουμε εστονική μετάφραση των τροπολογιών. Ζητώ συγγνώμη που παρενέβηνα, αλλά έπρεπε να εκφράσω αυτήν την ανησυχία μου. Μπορώ να ζητήσω από τον Νούνο Τεχέιρα να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι είναι ότι οι προϋποθέσεις ε, ε, ε, με τις οποίες δούλεψα εγώ όσον αφορά την έκθεση αυτή ήταν οι καλύτερες δυνατές. Την Τρίτη ή την Τετάρτη έθεσα ερωτήματα στους συναδέλφους και ζήτησα μάλιστα τότε και μεγάλη συνεργασία και διάθεση συνεργασίας από τους συναδέλφους έτσι ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε ε, σήμερα. Γιατί είναι σημαντικό να ψηφίσουμε σήμερα, μα γιατί θα υπάρξει ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες ως ο Νούπο και επομένως εάν δεν ψηφίζαμε σήμερα εδώ δεν θα μπορούσαμε να, ψηφίσουμε ε, την έκθεση στην επόμενη Ολομέλεια και επομένως δεν θα είχε πλέον έννοια η ύπαρξη αυτής της έκθεσης. Ζήτησα λοιπόν ναι, τον μέγιστο βαθμό συνεργασίας από τους συναδέλφους. Χαίρομαι που μπορούμε να ψηφίσουμε σήμερα, αλλά ταυτοχρόνως κατανοώ απολύτως ε, την δυσκολία των συναδέλφων που δεν μπόρεσαν να δουλέψουν στη γλώσσα τους. Ελπίζω πάντως ότι αυτό το πρόβλημα ε, δεν θα μας ε, εμποδίσει να συνεχίσουμε. Και η κυρία Κρέλ και ο κύριος Πίβολ θέλει να μιλήσουν βεβαίως δεν θέλουμε επί της ουσίας συζήτηση, απλώς να αποσαφηνίσουμε λίγο την ε, κατάσταση. Θα προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Και οφείλω να ρωτήσω αν διαφωνεί κανείς με την ψηφοφορία. Ο κύριος Πίπερ, δεν κάνουμε συζήτηση αρχής τώρα, αλλά θα μπορούσε να είναι προηγούμενο. Εάν το δεχτούμε τώρα. Εγώ εκτιμώ πολύ το συνάδελφο Τεσέρα και γνωρίζω και τη χρονική πίεση ε, στην οποία έχει υποβληθεί. Αλλά έχουμε μια έκθεση και πρέπει να κάνουμε τροπολογίες στα γαλλικά. Την άλλη φορά, εμείς είμαστε Γερμανοί, θα ζητήσουμε στα γερμανικά. Είναι μία από τις τρεις ε, γλώσσες εργασίας. Ε, τι είναι αυτό, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λέει η γραμματεία της Επιτροπής ότι υπάρχει αγγλική μετάφραση μεν, αλλά δεν εγγυόμαστε τίποτα. Ε, δεν μπορούμε να εργαζόμαστε έτσι. Αν είναι έκθεση πρωτοβουλίας, εντάξει. Αλλά αν είναι νομοθετικού περιεχομένου, ε, θα πρέπει να είναι πάντα πεντακάθαρη ε, η μετάφραση και να εμένουμε σε αυτήν. Αλλιώς δεν χάνουμε το καιρό μας κιόλας. Ε. Αν θέλετε να το αφήσουμε να περάσει αυτό τώρα ως εξαίρεση, αλλά κατά τα άλλα να μην αποτελέσει προηγούμενο και να έχουμε πάντα σωστές και καλές μεταφράσεις. Ευχαριστώ. Η πρόταση λοιπόν είναι να μην θεωρηθεί προηγούμενο, έτσι. Ε, όλα αυτά που αναφέρετε και εκφράσατε την απογοήτευσή σας να μην αποτελέσει παράδειγμα η προηγούμενο για το μέλλον. Καταλαβαίνω την πρόθεση κυρία Κλέρ. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον Μάρκους Πίπερ. Και εγώ το βρήκα λίγο δύσκολο, διότι οι σκιώδεις συγητές καταλαβαίνουν γαλλικά, αλλά οι συντονιστές λιγότερο. Τουλάχιστον εγώ τα γαλλικά μου δεν είναι και τόσο καλά για να καταλάβω αν οι συμβαστικέ τροπολογίες είναι εντάξει ή όχι. Και στην αρχή δεν είχα καταλάβει ότι πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί η πρότασή μας πριν την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το συζητήσαμε στην πολιτική μας ομάδα, λέγοντας ότι κανονικά δεν μπορεί το Κοινοβούλιο να λειτουργεί έτσι. Γιατί εμεί οι ίδιοι υποτιμούμε τον εαυτό μας και δείχνουμε ότι εντάξει μωρέ και τι έγινε. Ε, όχι. Αυτό δεν έχει να κάνει με το αν έχουμε καλές ή κακές σχέσεις με τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες. Και όταν ε, ζήτησα εγώ κάποια στιγμή αναβολή τη ψηφοφορία, βγαίνουν και λένε ότι οι σοσιαλιστέ και οι δημοκράτε είναι κατά των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών. Σε καμία περίπτωση. Πρέπει να ξέρω όμω τι αποφασίζω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η διαδικασία και οι τελευταίε αλλαγέ ε, για τι συμβαστικέ τροπολογίε έφτασαν σήμερα το πρωί στι 9. Και είχαμε δυσκολίες να φέρουμε στις 10 τον κατάλογο ψηφοφορίας που είναι και περίπλοκος πολύ. Θα πρέπει να ψηφίσουμε αργά και προσεκτικά γιατί έχει προβλήματα ο κατάλογος. Πραγματικά να θεωρηθεί απόλυτη εξαίρεση, να μην το ξαναζήσω παρακαλώ την παρούσα κοινοβουλευτική θητεία. Madame please. Κυρία Ναι. Εξ όσων γνωρίζω εγώ, είχε εκφραστεί επιθυμία να αναβληθεί η ψηφοφορία. Και τελευταία στιγμή μπήκε στην ημερήσια διάταξη. Και ιδιαίτερα ο κατάλογος ψηφοφορίας έφτασε σήμερα. Ο τελευταίος, με τις τελευταίες συμβαστικές προτάσεις που μόλις καταλήξαμε. Εγώ θα πρότεινα αναβολή της ψηφοφορίας. Γιατί στην αρχή οι ηγητές αυτό είχαν συμφωνήσει. Ακριβώς γιατί δεν είχαν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσεις και συζητήσεις. Ζητώ επισήμως αναβολή της ψηφοφορίας. Λαμπερ Φανίστεροι. Πρόεδρε, ο καθένας ε, και πολλοί είπαν ότι δεν είναι αυτή η μέθοδος και συμφωνώ. Θα ήθελα να πω το εξής ε, που ήταν καθοριστικό για μας. Είμαστε τώρα στην προετοιμασία των νομοθετικών προτάσεων. Ε, πρώτο αυτό. Δεύτερο, αυτή τη θητεία μία φορά, μόνο μία φορά, κάνουμε εμεί έγγραφο για τι ιδιαίτερα απομακρυσμένε περιφέρειες και είναι το παρόν και γνωρίζουμε ότι θα έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο και θα κάνει ανακοίνωση για τη δική του πολιτική επί τη ουσία και θα πρέπει να βασίζεται και στο δικό μα κείμενο. Και είναι και ένα νέο πλαίσιο με τη στρατηγική του 2020. Γι' αυτό το λόγο το είπαμε και στους συντονιστές Ζητώ να ψηφίσουμε και απευθύνω έκκληση στους ενδιαφερομένους. Τον Απρίλιο θα πάει στην Ολομέλεια και εμείς ως Κοινοβούλιο θα έχουμε το δικό μας όραμα, τη δική μας πρόταση και θα την έχουμε καταθέσει. Ένα μισή χρόνο νομίζω κρατάει αυτή η ιστορία και θα πρέπει να τελειώνει κάπου. Δεν ξέρω, κυρία Σρότερ λέει αναβολή της ψηφοφορίας. Εγώ κοίταξα το περιεχόμενο και την ουσία. Αν θέλετε να το ψηφίσουμε αυτό, αυτό είναι θέμα των πολιτικών ομάδων, αλλά γι' αυτό βιαζόμαστε και την περασμένη Τετάρτη είπαμε ας προσπαθήσουμε να το βάλουμε στη μερίσια διάταξη για να παίξει και ρόλο στη διαδικασία αυτή πριν την ανακοίνωση του Μαΐου και να μην έχουμε ένα έγγραφο το οποίο θα έρθει κατόπιν εορτής και τι να το κάνουμε. Αυτά. Ε, ο κύριος Γκουτμάνης τελευταίος είσαι ε, ομιλητής. Και εγώ ζητώ από όλους να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία για ένα πολύ απλό λόγο. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμού ε, εμείς ψηφίσαμε για την έκθεση αυτή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση γιατί οι περικοπές είναι πάρα πολύ μεγάλες φτάν, τη γνωμοδότηση αυτή της, της Επιτροπής ε, και ε, λόγω των υψηλών περικοπών ήταν πάρα πολύ σφιχτή η κατάσταση. Όμως αυτή την Πέμπτη θα έχουμε συζήτηση για το σύνολο του προπολογισμού, δηλαδή πόσα λεφτά θα πάρουμε. Και επομένως ε, είναι σημαντικό να δούμε αν θα πάμε στο συν 5% ή στο 3,16% που προτείνει η Επιτροπή και ελπίζω να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με μια συνολική περικοπή 10% στο συνολικό προϋπολογισμό. Μας απασχολούν πάρα πολύ όλα αυτά ε, και πώς είναι δυνατόν λοιπόν να ξεχάσουμε αυτές τις ιδιαίτερα προκριμένες ε, περιφέρειες και ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν αυτοί που ασχολούνται με τον προϋπολογισμό τη γνωμοδότησή μας γιατί διαφορετικά ε, τι θα γίνει. Θα προσπαθήσουν ε, ε, να μελετήσουν το θέμα και τα πόσα χρήματα θα δεσμευτούν χωρίς όμως να ξέρουν ακριβώς ποια είναι η άποψή μας. Ναι, κοιτάξτε, εγώ είναι γεγονός ότι δεν καταλαβαίνω καλά τα γαλλικά αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρξαν και πολλοί συμβιβασμοί άρα οι υπεύθυνοι και οι συντονιστές μας κάνανε συμβιβασμούς Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούσαμε και τον εισηγητή και τους ε, συναδέλφους που έχουν ε, ε, την άποψη ότι όντως υπάρχουν δυσκολίες και ότι ήταν τέλος πάντων προβληματική και ανησυχητική κατά την άποψή τους όλη αυτή η δύσκολη διαδικασία. Λέμε ότι εκπροσωπούμε εδώ μια επιτροπή και ότι και ο κανονισμός 156.6 ε, αναφέρει ότι θα πρέπει να αναβληθεί ε, η ψηφοφορία ε, μονάχα εάν, εάν υπάρξουν γλωσσικοί λόγοι ε, αλλά όμως ε, η, η συνάδελφος η οποία αναφέρθηκε στα γλωσσικά προβλήματα ε, δεν ζήτησε αναβολή της ψηφοφορίας. Επομένως δεν έχουμε επίσημο αίτημα για αναβολή λόγω γλωσσικών προβλημάτων. Εν πάση περιπτώσει... Ε, ε, συμφωνούμε ότι έχουμε δεσμευτεί όλοι, δηλαδή έχουν δεσμευτεί όλοι οι πολιτικοί συντονιστές καθώς επίσης ε, και όλοι οι πολιτικοί, τον, πολιτικοί συντονιστές των πολιτικών ομάδων έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν στην ψηφοφορία. Εν πάση περιπτώσει τώρα θα πρέπει να αποφασίσουμε είτε θα αναβάλουμε την ψηφοφορία λόγω γνωστικών προβλημάτων είτε θα προχωρήσουμε. Δεν βλέπω να επιμένει κανείς την αναβολή λόγω γλωσσικών προβλημάτων, επομένως... Προχωρούμε με την ψηφοφορία. Συμβιβασμό 6. Συμβιβασμός 6 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7 υπέρ Αγαπητοί συνάδελφοι, να σηκώνετε τα χέρια σας να βλέπω τι γίνεται. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ο κύριος Τυρολή. Χωρίς μικρόφωνο. Προφορική τροπολογία για το συμβιβασμό 7. Okay, so you're welcome to read, yeah. Α, ναι, να το διαβάσετε λαμβάνοντας υπόψη ότι ε, μπορεί μια ιδιαίτερα ότι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ε, ε, καταφέρει τους στόχους, να επιτύχει τους στόχους σε μια ιδιαίτερα απομαξιμένη περιφέρεια κτλ. κτλ. Ε, είναι κανείς κατά αυτής της προφορικής τροπολογίας. Όχι, επομένως ε, ψηφίζουμε ε, την, την, το συμβασμό 7 με αυτήν την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 76 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 87 υπέρ. 85, συγγνώμη. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 9 υπέρ. Ε, κύριε Τυρολή... Χωρίς μικρόφωνο, κύριο Στυριλίου. Ανησυχεί διότι η βρικοδότηση η οποία αρχικά ε, προτίθεται να καλύψει ε, το, τα ε, ιδιαίτερα προβλήματα αυτών των περιοχών. Θα ήθελα να πούμε αντί για αυτών των περιοχών να αναφερθούμε σε ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές και περιοχές με λίγο πληθυσμό. Είναι κανείς κατά, όχι, επομένως ψηφίζουμε το Συμβασμό 9 με αυτή την προφορική τροπολογία του κ. Τυρολία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ κατά. Τροπολογία 94 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεν θα ψηφίσουμε το 93. Το 93 έχει μπει στον ε, συμβασμό 8, λέει η Πρόεδρος. Σήμερα το πρωί εστάλει μία τροποποιημένη λίστα, ένας τροποποιημένος κατάλογος ε, ε, ψηφοφορίας.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 υπήρχε ένα τεχνικό λάθος, υπήρχε ένα τεχνικό λάθος ε, στη, στον κατάλογο και η κυρία Καρβάλιο τον διόρθωσε, αλλά δεν άλλαξε καθόλου η ουσία. Ήταν μια τεχνική διόρθωση και επομένως μπορούν και όσοι εμφιβάλλουν ε, να το δουν με την Κάρλα μετά την ε, ψηφοφορία. ψηφίσαμε την 94 και τώρα ψηφίζουμε την 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 114 με προφορική τροπολογία. Είναι κανείς κατά της προφορικής τροπολογίας, όχι. Επομένως ψηφίζουμε με την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, συμβιβασμός 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 127 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 19α είναι η 67, 92 και 152 ε, υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Εκατόν δεύτερο τμήμα, 112 δεύτερο τμήμα υπέρ, Ε, πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Τροπολογία 112, δεύτερο τμήμα, ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχιετή ψηφοφορία. Πέρας, απορρίπτεται. 18 υπέρ 21 ψήφοι κατά, άρα απορρίπτεται. Επομένως, περνούμε στην τροπολογία 158 υπέρ. Κατά υπέρ, υπέρ, υπέρ της 158. Κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 169, 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ κατά θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για το 171. The vote is open, the vote is moving, moving, closed I think. It's adopted. Εγκρίνεται 24 ψήφοι υπέρ 15 κατά. Ε, συμβασμός 22. Ε, Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Dear colleagues, there is a proposal. There is a proposal now that except for amendment. Λοιπόν, εκτός από την τροπολογία 4, όλες οι άλλες διαγραφές ε, ισχύουν. Ο εισηγητής λοιπόν προτείνει να διαγράψουμε τα πάντα εκτός από την 4. Εάν συμφωνείτε λοιπόν θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε ένα μπλοκ εκτός από την τροπολογία 4. Από το 1 μέχρι το 44 εκτός από το 4. Από το 45 μέχρι εκτός από το 4. Είπε κάποιος όχι. Δεν ακούν οι διερμηνείς δυστυχώς. Α, θέλετε τις τροπολογίες 2 και 4 χωριστά και επομένως από τη 1 μέχρι τη 45 on block. Ε, θα ψηφίσουμε on block πρώτα από τη 1 μέχρι τη 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εκτιμώντας τώρα, συμβιβασμός 1 ε, των εκτιμώντας υπέρ κατά αποχές Έχουμε προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε συμβιβασμό 2 επί των αιτιολογικών σκέψεων. Θέλετε κάτι να πείτε? Όχι. Συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβασμός 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβασμός 4 κατά ε, αποχές εγκρίνεται, συμβιβασμός 5 ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 62 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τώρα οι προτάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, ε, πρόταση 1, 4 λοιπόν, υπέρ, στην 4 πηγαίνουμε, υπέρ, κατά, Αποχές. εγκρίνεται, 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην 6, ναι, ε, πρόταση 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 8 καταπίπτει, επομένως τώρα περνάμε στις προτάσεις της Ήτρε. Πρόταση 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται υπαριθμών 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε τώρα την τελική ψηφοφορία. Θα γίνει ε, με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, υπάρχει ένας επιπλέον από την σοσιαλιστική ομάδα. Ένας επιπλέον. Ε, Επομένω, εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία 36 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, 4 αποχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όπως είχαμε συμφωνήσει, θα βγάλουμε από αυτά τα συμπεράσματά μας και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, αν θέλετε, στους συντονιστές για το τι θα κάνουμε σε τέτοιες Ε, Ερχόμαστε στο σημείο 12. Ο Γιάννη Όλμπερτ έχει το λόγο. Ξέρεις, είναι το θέμα σου. Μία ώρα και 22 ακριβώς λεπτά έχουμε για τρεις εκθέσεις. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και της Ρίκα Μάνερ για το ETC, για την εδαφική συνεργασία. Και έχουμε και τους συναδέλφους από την Επιτροπή Περιφερειών. Και θα τους παρακαλέσω να είναι όσο γίνεται πιο σύντομοι να μας διαβάζουν τις εκθέσεις τους, να μας τις παρουσιάζουν ε, με τρόπο ώστε να έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Είναι εδώ ο Μίχαλ Σνάιντερ, ελπίζω να είναι παρόν. Κάντε λίγο ησυχία για να ακούσουμε ήρεμα ε, τον ομιλητή μας θα συζητήσουμε σημαντικά θέματα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ακούμε πρώτα την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών και τον εισηγητή κύριο Μιχάλ Σνάιντερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Δεν είμαι πρώτη φορά εδώ. Ε, χαίρομαι όταν κάνουμε εντατική ανταλλαγή απόψεων. Μαθαίνω πάντα πάρα πολλά. Κοτέρ λέγεται η αρμόδια επιτροπή μας. Πριν από δύο εβδομάδες εγκρίναμε γνωμοδότηση για τον κανονισμό ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στην ωραία πόλη της Λισαβόνος. Το Μάιο θα έρθει στην Ολομέλειά μας και θα ήθελα πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω ορισμένα ε, σημαντικά και κεντρικά θέματα για τη γνωμοδότηση αυτή. Για λόγους χρονικούς θα αφήσω στην άκρη ε, τους γενικούς επένους του κανονισμού και τα λοιπά. Ε, αξιολογούμε θετικά ε, καταρχήν τον κανονισμό, αυτό το προεξοφλώ και δεν θα επεκταθώ, θα μπω στις λεπτομέρειες. Άρθρο 3 του κανονισμού. Πρόκειται για τους τομείς παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εμείς εδώ θεωρούμε ότι οι τομείς παρέμβαση που αναγράφονται σε αυτόν τον κατάλογο προσφέρονται και για την υλοποίηση των στόχων ε, της πολιτικής συνοχής που είναι κατοχυρωμένη στη συνθήκη αλλά και για τη στρατηγική του 2020. Αυτά τα δύο μπορούν να επιτευχθούν. Ωστόσο, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή ότι σε αντίθεση με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε ανεπτυγμένες περιφέρειες ε, μπορεί να χρειαστεί να επενδύσουν σε υποδομές για παροχή υπηρεσιών ε, κοινή ωφέλεια ε, στην επικοινωνία, τεχνολογία και στις συγκοινωνίες. Δηλαδή, όχι στις πιο αδύναμες περιφέρειες, αλλά και στις πιο ανεπτυγμένες. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα τέτοιων επενδύσεων. Επίσης, θεωρούμε ότι η υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων με άμεσες ε, ενισχύσεις επενδυτικές μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν αρκεί για να φτάσουμε στους στόχους της βιομηχανικής πολιτικής τα ε, ε, χρόνια της παγκοσμιοποίησης. Θεωρούμε ότι και στο μέλλον θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επενδυτικής ενίσχυσης και μεγάλων εταιριών να μην καταργηθεί αυτή η δυνατότητα. Οι πολλές περιφέρειες και το γνωρίζουν οι περιφέρειες και οι Επίτροποι Περιφερειών. Σε πολλές περιφέρειες οι μεγάλες εταιρείες παίζουν ρόλο διαρθρωτικής πολιτικής. Πολύ μεγάλες επιχειρήσεις αναθέτουν ε, σε υπεργολάβους, σε μικρότερες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες και οι, μεγάλες ε, εταιρείες όταν δέχονται ενισχύσεις έμεσα ενισχύουν και τις μικρές. Άρα λοιπόν ε, οι παραγωγικές πάντα επενδύσεις θα πρέπει να ενισχύονται όχι μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε μεγαλύτερες για τη σύσταση, διεύρυνση ή διαφοροποίηση εργοστασίων ή ριζική αλλαγή μεθόδων για παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών που δημιουργούν και διατηρούν αηφόρες θέσεις απασχόλησης και βιώσιμες. Αν δούμε λοιπόν τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως το θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μειώσει τις ενισχύσεις και τις επενδύσεις σε εταιρείε ε, και μιλά μόνο για startups, για νέες εταιρείε, ε, τότε αυτό δεν ανταποκρίνεται ε, στις καταστάσεις και στις προκλήσεις των περιφερειών. Και σε ό,τι αφορά λοιπόν του τομείς παρέμβασης θεωρούμε ότι στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί για ε, τα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα. Δηλαδή να, να, να ενισχύουμε μόνο τα δημόσια κέντρα, θα μπορούσαν να ενισχύονται και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα. Και ιδιαίτερα κοινά ερευνητικά προγράμματα ιδιωτικά ιδιωτών και δημοσίου. Δηλαδή ε, ερευνητικά κέντρα που μπορεί να είναι ιδιωτικά και να συνεργάζονται με πανεπιστήμια και άλλα τέτοια τεχνολογικά Ινστιτούτα. Όλα αυτά για το άρθρο 3. Έρχομαι στο 4. Η θεματική συγκέντρωση. Ε, φαντάζομαι ότι είναι το θέμα κλειδί για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και χρειάζεται εξήγηση. Εμείς έχουμε πολύ επικριτική θέση για το άρθρο 4. Θεωρούμε μεν ότι καταρχήν ε, θα πρέπει να υπάρχει θεματική συγκέντρωση Δηλαδή σε θεματικούς στόχους έχει νόημα κάπου να συγκεντρώνεται κανείς και είναι σκόπιμο αυτό, αλλά εμείς απορρίπτουμε την κεντρική απόφαση και τον επιμερισμό των πόρων για τις θεματικές ε, προτεραιότητες. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται στην περιφέρεια. Ε, ε, εκεί είναι το κατάλληλο επίπεδο, όχι το κεντρικό, για να αποφασίζεται η συγκέντρωση των στόχων και των προτεραιοτήτων. Το άρθρο 4 κάνει κάποιες προτάσεις αλλά δεν επιτρέπεται αυτό να ορίζεται, να υπαγορεύεται από το κέντρο. Οι περιφέρειες να έχουν λόγο σε εταιρική σχέση. Και οι οργανισμοί τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης έχουν αρμοδιότητες και θα πρέπει να συμμετέχουν από τον προγραμματισμό, να λένε ποια είναι η στρατηγική ανάπτυξη περιφέρειας, αυτόνομα, ε, με αυτοτέλεια, με ε, μεμονωμένες ε, και προτεραιότητες και με τη στρατηγική για το 2020 από την πλευρά τους, όχι να τους θα υπαγορεύουν αυτά τα κράτη. Άρα εμείς καταλήγουμε στο συμπέρασμα να απαλληφθεί η παράγραφος 4 σχεδόν στο σύνολό της, ε, με εξαίρεση την πρώτη φράση. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ αυστηρή και άκαμπτη θέση, το συζήτησα με τον Επίτροπο Χάν και έκανα μια προσφορά να προσπαθήσουμε για την Ολομέλεια του Μαΐου να βρούμε μια συμβαστική λύση Βλέπω κάποια στοιχεία συμβιβασμού στις προτάσεις. Το 80% που είναι πολύ υψηλή, ε, υψηλός ποσοστό για τις αναπτυγμένες περιφέρειες, να υπάρχει μια ευελιξία και για το κοινωνικό ταμείο και οι δυνατότητες χρηματοδότησης του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης να μην περιορίζονται στις ε, μικρομεσαίες και να μπορούν να χρηματοδοτούνται και κάποιες άλλες υποδομές πέρα από όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτο τελευταίο, το άρθρο 7, αηφόρος αστική ανάπτυξη. Και εδώ θεωρούμε ότι θα πρέπει να τα ορίζουν αυτά λιγότερο τα κράτη σε κεντρικό επίπεδο για το πώς θα αναπτύσσεται μια πόλη ε, και πόσο μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη και οι περιφέρειες να έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια των ε, ΕΣΠΑ να βλέπουν πώς θα αναπτύσσουν τις πόλεις τους. Ένα 5% ως προσανατολισμό. Δεν είναι τελείως απορριπταίο. Αυτό που είναι για μας απορριπταίο είναι να ορίζει κάποιος κεντρικά τι θα κάνουν οι πόλεις αποκεντρωμένα και στα πλαίσια των εταιρικών σχέσεων και συμβάσεων θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η συγκέντρωση δεν πρέπει να αφορά μόνο αστικές ε, περιοχές αλλά και τις λεγόμενες περιαστικές ή μη υπαίθριες, υπαίθριες και εκεί να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Σε σχέση με όλα αυτά θεωρούμε ότι ο κατάλογος που προβλέπεται για τις πόλεις δεν είναι σκόπιμος. Θα πρέπει να ε, υπάρχει μια ανοιχτή προσέγγιση, δηλαδή να, όχι ένας κλειστός κατάλογος, ε, να υπάρχει αν θέλετε κατάλογο, ενδεικτικός κατάλογος πόλεων. Σε σχέση με την αστική ανάπτυξη και οι ε, ενσωματωμένες εδαφικές επενδύσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 99 του Γενικού Κανονισμού, και πάλι δεν θέλουμε τα μέτρα αυτά να είναι δεσμευτικά, να είναι επιλογή Καλώς, Οι διοικητικές ε, υπηρεσίες που φέρουν την ευθύνη στις περιφέρειες για τα οικονομικά θα πρέπει να συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές και να λαμβάνουν υπόψη τις τεχνικές και θεσμικές δυνατότητες και να μπορούν να αποφασίζουν από μόνες τους ε, πώς θα αναθέτουν και σε ποιο βαθμό ε, τις εξουσίες. Το άρθρο 8, το Φόρουμ για την Ανάπτυξη των Πόλεων δεν κατανοούμε για ποιο λόγο να χρειάζεται ένα τέτοιο φόρουμ. Έχουμε ένα θαυμάσιο πρόγραμμα που ονομάζεται URB Act. Οι συμμετέχοντες όλοι το εκθιάζουν. Γιατί να έχουμε τώρα νέο φόρουμ. Υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό όργανο που εκπροσωπεί και πόλεις και ονομάζεται Επιτροπή των Περιφερειών. Δεν εκπροσωπεί μόνο τις περιφέρειες αλλά και δήμους. Έχουμε ε, δημάρχους τύπου Λισαβόνας, Φραγκφούρτης και τέτοια Μπορεί και η Επιτροπή Περιφερειών να συνεργάζεται και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα είμαστε στη διάθεσή σας για να κάνουμε πολλά χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστό φόρουμ για τις πόλεις. Τελευταίο. Στο άρθρο 10 της πρότασης κανονισμού αναφέρονται κάποιες ρυθμίσεις για ε, περιφέρειες που έχουν μειονεκτήματα δημογραφικά όσο και γεωγραφικά Έκανα εγώ μια ακρόαση ως εισηγητής για τα δημογραφικά αυτά προβλήματα σε άλλες περιφέρειες από αυτές που μας απασχολούν μέχρι τώρα. Και φάνηκε ότι υπάρχουν μια σειρά ευρωπαϊκών περιφερειών που υπάρχουν δημογραφικά προβλήματα και διαδικασίες. Μειώνει το πληθυσμός δηλαδή. Και αυτό έχει πολύ μεγάλες ανητικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη αυτών των περιφερειών. Κατά την άποψή μας θα πρέπει να εξασφαλιστεί στα πλαίσια του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης να είμαστε έτοιμοι για νέες δημογραφικές προκλήσεις. Πέρα από τις κλασικές που βεβαίως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά υπάρχουν και νέες δημογραφικές προκλήσεις και χρειάζονται νέες απαντήσεις από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτά αυτή είναι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών. Αν σας ενδιαφέρει, την έχουμε και ε, κείμενο, την έχουμε φέρει μαζί μας. Συγκεκριμένες προτάσεις για κάθε άρθρο. Κατανοώ ότι υπάρχουν προβλήματα με τη διαδικασία αυτή, αλλά δυστυχώς αυτή είναι, δεν έχουμε άλλη. Ε, σας παρακαλώ, κοιτάξτε το έγγραφό μας και κύριε Όρμπρεχτ, ελπίζω να παραμείνουμε σε στενή επαφή για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Όλμπριχτ. Ευχαριστώ κύριο Όλμπριχτ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ σαφή πρότασή του και ε, κάναμε ανταλλαγές απόψεων και ε, όντως ε, τώρα κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Ε, σχετικά με τις λεπτομέρειες. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία ανέφερε ο εισηγητής και θεωρούμε ότι είναι βασικά για την έκθεσή μας στο Κοινοβούλιο. Καταρχήν είναι το θέμα του άρθρου 3 σχετικά με την εμβέλεια της στηρίξεως που έχει και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Το αρνητικό είναι ότι ε, όσον αφορά τις ε, επενδύσεις ε, υποδομής ακούσαμε ότι Είμαστε από την Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για τις κλιματολογικές αλλαγές, ότι ε, υπάρχει μία δυνατότητα και μπορούμε να δούμε ε, ποια είναι η, ποιο είναι το θέμα σχετικά με το ICTS, με την European Transport Facility, το μέσον για τις μεταφορές. Αλλά βλέπω εδώ ότι επαναλαμβάνεται η ισχύουσα κατάσταση και ουσιαστικά πρόκειται για τις ε, υπηρεσίες υποδομές. Βλέπουμε λοιπόν ότι ό,τι υπάρχει και σήμερα <laughs> θα υπάρχει και αύριο. Οπότε έχουμε όλο και περισσότερες ενδείξεις από τις ανεπτυγμένες περιοχές ότι δεν έπρεπε να είμαστε τόσο αυστηροί δεν έπρεπε να απαγορεύσουμε τόσο σταθερά αυτές τις επενδύσεις. Η κατάσταση όμως αλλάζει. Υπάρχει μία περίοδος κρίσεως, κλιματολογικές αλλαγές και είναι όντως αναγκαίο να προχωρήσουμε χωρίς να κλείσουμε τελείως την πόρτα. Επίσης για τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει μία πλήρης απαγόρευση για τις ε, παραγωγικές ε, επενδύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά τις ε, παραμεθόριες ακραίες περιοχές οι οποίες συνεργάζονται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν λοιπόν οι μεγάλες επιχειρήσεις αποκλειστούν από το παραγωγικό έργο τότε ε, ε, με επισκέφθηκαν ε, οι υπεύθυνοι για την παραγωγή στην περιφέρεια και μου είπαν ότι μεγάλες παγκόσμιες επιχειρήσεις μπορούν να κινηθούν και στις ακραίες περιοχές και δεν θα έπρεπε να αποκλείονται. Προτείνω λοιπόν να πούμε ότι οι μεγάλες εταιρείες, ε, αυτές οι οποίες συμμετέχουν στις ε, ε, παραγωγικές διαδικασίες, είναι σε συνδυασμό με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν πρέπει να αποκλείονται. Πρέπει δηλαδή να βρεθεί κάποιος τρόπος για συμβιβασμό, διότι σας υπενθυμίζω ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν αποκλείονται από πλευράς ε, στηρίξεως ε, εις ε, την ε, ε, ε, στο χώρο αυτό. Αυτό είναι το ένα στοιχείο, δεν πρέπει να τις αποκλείσουμε. Δεύτερον, ο εισηγητής προτείνει να διαγράψουμε τελείως το άρθρο 4, αλλά υπάρχει συναπόφαση με το Συμβούλιο και το Συμβούλιο μας ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει ακραία θέση σχετικά με το άρθρο αυτό, δηλαδή τα περισσότερα κράτη-μέλη συμφωνούν. Δεν πρέπει να υπάρξει αυτόματο συγκέντρωση Οπότε πρέπει να δούμε ή να αλλάξουμε το ποσοστό από 80 σε 60 σε 70 δηλαδή να αλλάξουμε τα ποσοστά ή να προτείνουμε να υπάρξει μία συγκέντρωση αλλά θα πρέπει οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα υπάρχει η συγκέντρωση να ε, αποφασιστούν από τους υπευθύνους, αν θα είναι το 153 ή το 158. Δηλαδή οι, θεματικές, ε, οι θεματικοί στόχοι δεν πρέπει να είναι τόσο αυστηροί. Ε, όσον αφορά την ενεργειακή ε, αποτελεσματικότητα επίσης. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι μία τέτοια πρόταση θα είναι πλήρως αποδεκτή αλλά 80% με αποκλεισμό της μεταφοράς της πόλης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Επίσης πόσο αναφέρομαι ή στις μεταφορές της πόλης με χαμηλή εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή ε, αποκλείεται. Οπότε το άρθρο 4 είναι πολύ σημαντικό. Σχετικά με το άρθρο 5, το συζητήσαμε χθε. Σας υπενθυμίζω την πρόταση μου η οποία είναι καταρχήν όσον αφορά τη συμφωνία συνεργασίας που προβλέπεται στις γενικές ρυθμίσεις και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ήταν ε, πολύ αυστηρή στη συνθήκη αυτή και ε, ακολουθώ την ίδια γραμμή. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να αφαιρεθεί τελείως από τον κατάλογο και να μην υπάρχει ενδεικτικός κατάλογος διότι αυτός μπορεί να σημαίνει πολλά. Προτείνω λοιπόν να διαγραφεί τελείω και να μιλάμε για κριτήρια, δηλαδή έναν κατάλογο κριτηρίων. Ε, υπάρχει μια συγκεκριμένη δράση για το 5% και η δράση αυτή του 5% σύμφωνα με την πρότασή μου προς την Επιτροπή θα πρέπει να αναφέρεται εις τα λειτουργικά θέματα που θα αποφασίζεται ε, οι περιοχές αυτές, οι λειτουργικές περιοχές να ρυθμιστούν σε εθνικό επίπεδο είτε μικρές πόλεις ή ένα μείγμα περιοχών και κάποιο συνδυασμός με το περιβάλλον γύρω από τις πόλεις. Ε, και κατά τη δικιά μου άποψη και δεν έχω εδώ αλλάξει τις απόψεις μου ακόμη και μετά από τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προτείνω στην έκθεσή μου τη δυνατότητα για τις πόλεις να μπορέσουν να καταλήξουν εις ε, το χώρο δηλαδή να υπάρχει μία, ή ένας ειδικός τρόπος αναθέσεως διότι αλλού υπάρχει πλήρης ανάθεση και αλλού υπάρχει μερική ανάθεση, δηλαδή βάση επιλογής προγραμμάτων κτλ. Εκεί αναφέρεται αυτό το 5%. Και βεβαίως, ε, λογικά, σύμφωνο ότι εάν εγκαταλείψουμε την, ε, ε, τον κατάλογο θα πρέπει να εγκαταλείψουμε και την πλατφόρμα διότι η πλατφόρμα υπάρχει για τον κατάλογο. Ο τρόπος αξιολογήσεως, παρακολουθήσεως και τα λοιπά μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είτε από τις ισχύουσες ε, δομές είτε από το ταμείο. Δηλαδή το νομικό αυτό κείμενο που δεν είναι μία επεξήγηση, είναι ένα νομικό ε, κείμενο, δεν πρέπει να δημιουργήσει μία νέα πλατφόρμα. Κατάλαβα τι εξηγήσατε, αλλά θέλω να πω ότι εδώ στο έγγραφο έχουμε μία θετική αξιολόγηση των δικτών ε, και εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν ε, έχω θετική άποψη για τους δείκτες πιστεύω ότι είναι υπερβολικά ε, γενική, ασαφής και δεν αναφέρονται στις συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες θα ήθελα λοιπόν περισσότερη σαφήνεια στους δείκτες γιατί οι δείκτες αυτοί προτείνονται σε διάφορους τομείς οι οποίοι όμως διαφέρουν από αυτούς που περιέχονται στον κανονισμό. Ο κανονισμός δεν αναφέρεται στην πολιτική των πόλεων ενώ έχουμε δίκτυα τα τετραγωνικά ε, που αναφέρεται στις πόλεις. Επίσης όσον αφορά τις ε, ε, πόλεις, ε, τους χώρους των πόλεων. Τι εννοείται με αυτό, όλα αυτά θα ήθελα να διευκρινιστούν. Προτού να ζητήσω την ε, κυρία Βεσφάλεν και την κυρία Σάντσε Σμιτ, θέλω να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με τις μικρές ε, και τις μεγάλες επιχειρήσεις, διότι δεν ισχύει ότι δεν ε, επωφελούνται στις περιοχές συνοχής, αλλά υπό κάποιον όρο, δηλαδή για να μην υπάρξουν μετακινήσεις ε, ε, επιχειρήσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρέπει ε, να δούμε εάν μετακινούνται επιχειρήσεις αυτό να μην οφείλεται εις το ευθυνότερο εργατικό δυναμικό και έχει τεθεί ένα ποσοστό στα κράτη-μέλη δηλαδή μέχρι 60-70% θα πρέπει να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μετά ξεκινούν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Οπότε πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, ιδίως στον τομέα των καινοτομιών. Ε, οι μικρές επιχειρήσεις βοηθούν τις μεγάλες να προσχωρήσουν σε την αλυσίδα προμηθειών. Υπάρχει δηλαδή ε, κάποια προϋπόθεση η οποία, την οποία προτείνουμε. Η κυρία Βέσφαλεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σνάιντερ για τα σχόλιά σας και πρέπει να σας πω ότι ιδίω η συνάντηση μεταξύ του ε, ε, της Επιτροπής, μεταξύ Επιτροπής και Επιτροπής του Κοινοβουλίου για το περιβάλλον είναι μια πολύ ευτυχής ιδέα αλλά βλέπω επίσης ότι πιο πλούσιες περιοχές ουσιαστικά δεν επενδύουν όσο θα έπρεπε στις υποδομές ούτε στον τομέα του περιβάλλοντος και των μεταφορών και επικοινωνιών. Εγώ όταν εξετάζω την χώρα μου και κοιτάζω το θέμα της ευρυζωνικής επικοινωνίας ε, και το θέματα που συζητήθηκαν σήμερα δεν βλέπω μεγάλη πρόοδο. Η δημογραφία περιέχει και τον όρο δημοκρατία και σαν εισηγήτρια για την ε, Επιτροπή Περιφερειών για τις δημοκρατικές αλλαγές είναι ένα θέμα που με, πλή, με ενδιαφέρει πάρα πολύ και βλέπω ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη επέμβαση διότι δεν είναι δυνατόν η δημογραφία να αναφέρεται εν παρόδο εφόσον πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος ε, ήδη, ήδη επηρεάζει την κατάσταση εφόσον μειώνεται η πυκνότητα του πληθυσμού. Επίσης ε, πρέπει να αντιδράσουμε καλύτερα όσον αφορά τις ε, πιο μειονεκτικές περιοχές. Ε, ένα άλλο θέμα που εφήγει αλλά το οποίο επίσης με ενδιαφέρει είναι αυτό που σας προανέφερα. Και πιστεύουμε ότι η πρόθεση των πόλεων θα πρέπει να αναφέρεται ρητός και να επηρεάσει ε, το, την έκθεση. Το κατώτατο επίπεδο το 5% κατά τη γνώμη μου είναι καλό, δεν πρημοδοτεί τις ε, πόλεις ε, αλλά αφήνει πίσω την ύπεθρο όταν λάβει κανείς υπόψη πόσο αναπτύσσονται οι πόλεις. Αλλά η βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων θα πρέπει να διατίθεται σε όλες τις πόλεις, είτε είναι σε μια μητροπολιτική περιοχή, είτε είναι σε μια ευνοημένη περιφέρεια και είπαμε χθε ότι το άρθρο 7 δεν μπορεί να λειτουργήσει αποκλειστικά και πιστεύω ότι στην Επιτροπή αυτή θεωρούμε ότι ο κατάλογος είναι αναγκαίος. Τώρα, αν χρειαζόμαστε το φόρουμ των, της ανάπτυξης των ε, πόλεων ή όχι είναι κάτι που δεν μου έχει διευκρινιστεί. Διότι εχθέ ελέγχθη ότι υπάρχουν εναλλακτικέ λύσει, και τις ανέφερε και ο κύριος Όλμπριχτ Μόλι. Και υπάρχουν διάφορα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε, δηλαδή την πρόθεση των επιχειρήσεων, η οποία επίσης θα πρέπει να ακολουθήσει και επιπλέον ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση για να προωθηθούν οι επενδύσεις, διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και ε, η πιο σημαντική ε, στήριξη των εργαζομένων εργαζομένων στην Ευρώπη. Ε, ενώ είμαι πιο επιφυλακτική για τις μεγάλες επιχειρήσεις, διότι πιστεύω ότι ε, ε, έρευσαν ε, ε, έρευσαν χρηματοδοτήσεις προς τις μεγάλες αυτές επιχειρήσεις που δεν έπρεπε να στηριχθούν από τους Ευρωπαίους φορολογουμένους. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να ξανασυζητήσουμε το θέμα και θα πρέπει να επεξεργαστούμε και ορισμένους δείκτες. Και τέλος ε, και εμείς ανησυχούμε για, την, για το θέμα των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί διότι η ε, θεματική συγκέντρωση είναι σημαντική όπως είναι σημαντική και επικέντρωση στους στόχους του 2020 και στηρίζουμε τις διάφορες προτάσεις αλλά το Ταμείο αυτό θα πρέπει να ε, εξισορροπήσει ορισμένες ε, ανισότητες και αυτό αναφέρεται στο άρθρο 2 και θα πρέπει επίσης να συζητείτε. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί ε, ε, αλλά θα χρειαστεί μεγαλύτερη ευελιξία για τις ε, περιφέρειες διότι υπάρχουν περιφέρειες όπου το θέμα έχει προχωρήσει περισσότερο από άλλες. Όσον αφορά την Γερμανία πιστεύω ότι υπάρχει ε, υπερβολική συγκέντρωση και αυτό δημιουργεί δυσκολίες και θα παραμείνω εδώ για τα σχόλιά μου. Συνάδελφοι, έχω τρεις ε, ομιλητές για να τελειώσουμε με αυτή την έκθεση. Άλλος κανείς να κλείσω το κατάλογο. Μάλιστα. Uh, Μάλλον δεν θα μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα τα θέματα πριν τις 12 όσο προλάβουμε και μετά για το απόγευμα. Και η Ρίκα Μάνερ, σκιώδη συγγήτρια των φιλελευθέρων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή ε, τη Επιτροπή των Περιφερειών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εξαιρετική έκθεση που είμαι βεβαίω ότι θα μας χρησιμεύσει, θα μας ε, φανεί χρήσιμη. Ήταν πάρα πολύ σαφής ε, σε όσα μας είπε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό λοιπόν εντάχει θα αναφερθώ σε μερικά από τα κατά την άποψή μου σημεία κλειδιά. Όσον αφορά τώρα την χρήση της ε, χρηματοδότησης ε, για ε, υποδομές σχετικά με την χρήση τους δηλαδή σε πιο αναπτυγμένες περιοχές πιστεύω ότι είναι καλό. Όπως είπε και ο εισηγητής θα ήταν καλό να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την ευρωζωνικότητα ας πούμε <coughs> γιατί έτσι θα βελτιωθεί ε, και η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κάποιες περιοχές. Όσον αφορά τώρα τα δημογραφικά διακυβεύματα, συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε. Οπωσδήποτε θα πρέπει να ληφθούν καλύτερα υπόψη στις ε, μελλοντικές προγραμματικές περιόδους. Λοιπόν, συμφωνώ πολύ ε, με τον ε, κατάλογο ή τέλο πάντων με τα κριτήρια ε, όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις αυτές. Αλλά βεβαίως τα κριτήρια θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι διαφορές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει να αποφασίζονται και σε εθνικό επίπεδο. Συμφωνώ λοιπόν με τον εισηγητή που λέει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές περιοχές, οι διαφορετικές συνθήκες δηλαδή ε, στα κράτη-μέλη. Δεν είμαι ε, υπέρ αυτής της αστικής πλατφόρμας, urban platform, Δύο λόγια ήθελα να πω επίσης όσον αφορά τις ε, επενδυτικές προτεραιότητες. Ε, πρώτα απ' όλα μην ε, λησμονούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιφερική ανάπτυξη να μην λησμονούμε την καινοτομία και τις πλατφόρμες καινοτομίας. Θα πρέπει δε να στηρίζουμε τη δημιουργία τέτοιων πλατφορμών την, ε, την συνένωση σε κλάστερς, την ε, δυνατότητα ε, κοινής και συντονισμένης αντιμετώπισης της δυνατότητας οικοδόμησης δυνατοτήτων, τις αντισταθμίσεις με τρόπον ώστε να έχουμε ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών και με τρόπον ώστε να βοηθήσουμε και άλλους να έχουν πρόσβαση είστε ιδιωτική ή δημόσια χρηματοδότηση. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνούμε την ε, πραγματική ε, καινοτομία καθώς επίσης ε, και την κοινωνική δικτύωση και το ρόλο που μπορεί να παίξει στην καινοτομία. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, ε, βοηθηθεί η ικανότητα, η οικοδόμηση μάλλον ικανοτήτων για ε, ξεκίνημα νέων επιχειρήσεων που θα δώσει νέα ζωή στις περιφέρειες και βεβαίως θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Όσον αφορά τώρα τις διεθνείς διασυνδέσεις, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε ε, ε, δίκτυα και βεβαίως ε, σημαντική θα είναι και η ανάπτυξη των υπηρεσιών. Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε την έρευνα και την ανάπτυξη στο ίδιο πλαίσιο. Η οικονομία με χαμηλό διοξίδιο του άνθρακος. Βεβαίως συμφωνούμε και θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω επενδύσεις έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Ε, οπωσδήποτε εγώ είμαι υπέρ τέτοιων δραστηριοτήτων. Όσον αφορά δε το πόσα χρήματα θα πρέπει ε, να ε, βρούμε για τα, για, τις, ε, για τα έργα αυτά, ε, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα. Θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω για το θέμα αυτό. Έχουμε την πράσινη οικονομία, ας πούμε, την οικονομία η οποία θα βασίζεται σε όλο και λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα, αλλά ταυτοχρόνως θα πρέπει να βοηθήσουμε τη μεγαλύτερη επένδυση, άρα να υπάρχουν αντισταθμίσματα, αντισταθμίσεις οικονομικές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Ντελή. Εγώ συμμερίζομαι απολύτως ε, τα ερωτήματα και ανησυχίες ε, του συναδέλφου Όλμπριχ σχετικά με την χρησιμότητα αυτής της πλατφόρμας. Υπάρχει ένα πρόβλημα μεθοδολογίας κατά την άποψή μου. Έχουμε τον κατάλογο των πόλεων που δεν πρέπει να καθοριστεί χωρίς ε, προηγούμενο καθορισμό των ολοκληρωμένων στρατηγικών. Επομένως πρέπει να είμαστε συνεκτικοί όσον αφορά την ανάπτυξη και την αναπτυξιακή πολιτική των εδαφών μας και επομένως περισσότερο από ποτέ στη διαπραγματεύσεις με τα κράτη θα πρέπει να αναμειχθούν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Εγώ πιστεύω πίσω ότι θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη αναφορά στις ε, περιαστικές ε, ε, πλατφόρμες όπως το αναφέρει άρρωστη και η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της City of Tomorrow και κατά την άποψή μου αυτό θα πρέπει να φαίνεται σαφώς στον καθορισμό των ολοκληρωμένων στρατηγικών. Θα επανέλθω σε κάποια ερωτήματα. Κατά την άποψή μου, και πάντα αναφέρομαι στην ίδια πλατφόρμα, κυρίως δε την επιλεξιμότητα των πόλεων. Εάν το ίδιο το κράτος καταρτίζει τον κατάλογο των πόλεων ε, για τη δημιουργία τελικών σχέσεων που θα υλοποιήσουν ε, τις στρατηγικές αυτές, τις ολοκληρωμένες στρατηγικές, τότε το ΟΥΡΠΑΚ θα ε, εξαφανιστεί. Και για μένα αυτό είναι κακό, γιατί το Ουρμπακ είναι πολύ καλό εργαλείο. Επίσης, όσον αφορά τις ε, κατά προτεραιότητα επενδύσεις, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει και άλλωστε το κατανοεί απολύτως και η Επιτροπή των Περιφερειών ε, το ζήτημα της στέγασης ε, κυρίως δε το σύστημα της ενεργειακής έλλειψης βλέπουμε ότι ε, αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο, μια μεγάλη πρόκληση όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές και επομένως δημιουργία θέσεων εργασίας, ε, σταθερές αμοιβέ και ταυτόχρονη μείωση της της, ε, του ενεργειακού λογαριασμού, αυτό είναι ένα μεγάλο διακύβευμα. Επίσης, πώς θα μπορέσουμε να ε, βγάλουμε, να, να, να βγάλουμε αυτά τα όρια, τα φανταστικά που υπάρχουν γύρω από συγκεκριμένες γειτονιές και τι σημαίνει συγκεκριμένα όταν λέμε ότι θα επιδοτηθούν ή ε, χρήση μέσων ε, μαζικής μεταφοράς. Αυτό δεν είναι πολύ σαφές. Επίσης το άρθρο 4 κυρίως ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε το ποσοστό των αναπτυγμένων και κυρίως τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε αναπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες μεταβατικές. Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε να επιμείνω σε τρία σημεία για μία ακόμα φορά ε, να δοθεί η άδεια ε, για περαιτέρω δημιουργία υποδομών, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών ε, στις αναπτυγμένες περιφέρειες. Αυτό το λέει και το ζητάει και η Επιτροπή Περιφερειών και πολύ μεταξύ ημών. Δεύτερον, ε, να διευρυνθεί η επιλογή των επενδύσεων των επιλογμένων περιοχών πέραν των ε, τριών αναφερομένων, κυρίως όσον αφορά την ε, τεχνολογία και την επικοινωνία. Τρίτον, Φαίνεται ότι ο φτωχό συγγενή του κανονισμού είναι ο πολιτισμό. Δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη με τρόπο βέβαια στρατηγικό και συνεκτικό εμφανίζεται μονάχα στο άρθρο 6, αν δεν κάνω λάθος, προστασία και προώθηση της πολιτιστικής χειρονομιάς. Θα πρέπει οπωσδήποτε να διευρυνθεί η αναφορά αυτή. Επίσης έχουμε στο σημείο 15 ε, και μία μελέτη που θα καταδείξει τη σημασία του πολιτισμού. Η προώθηση του πολιτισμού και της ε, οικονομίας ε, του δημιουργικού τομέα νομίζω ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις διαρθωτικές αλλαγές. Η κυρία Κορνέλισεν. Κορνέλιαν, ευχαριστώ και την Επιτροπή Περιφερειών καταρχάς. Είναι σταρά τα λόγια και καλό είναι που κάνετε έτσι ακραίες προτάσεις και ριζικές προσφορές για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε. Έτσι γίνονται τα πράγματα και συμφωνούμε σε πολλά. Σύντομα και συνεχτικά βεβαίως θα πρέπει και αναπτυγμένες ε, περιφέρειες να δουν τις βασικές επενδύσεις τους να ενισχύονται και εμείς το υποστηρίζουμε, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες αυτό. Επόμενο θέμα. Μικρομεσαίες. Ε, να προσανατοριζόμαστε εκεί αποκλειστικά. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να διευρύνουμε αυτό το βήμα όντω. και να εντάξουμε και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκεί. Ιδιαίτερα ακριβώς σε σχέση με τις διαθρώσεις και τις δομές των μικρομεσαίων σε μια περιφέρεια. Γιατί υπάρχει σύνδεση μεγάλων επιχειρήσεων με μικρές της περιφέρειες. Δεν θα πρέπει να αποκλείονται από την προσπάθεια αυτή αυτό για τις εταιρείε. Όχι περιορισμό στα δημόσια ερευνητικά κέντρα. Θα πρέπει νομίζω να επανέλθουμε σε μια διατύπωση που έχουμε στον ισχύοντα κανονισμό που λέμε ότι ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα ιδιαίτερα όταν έχουν κοινά προγράμματα με ε, δημόσια κτλ. θα πρέπει να ενισχύονται. Τουλάχιστον να το προτείνουμε. Οι θεματικές συγκεντρώσεις τρεις στόχοι είναι πολύ περιορισμένο και πολύ στενό και αυθαίρετο, χωρίς αιτιολόγηση. Δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε. Σε όλες τις συζητήσεις πάγια επαναλαμβάνουμε ότι αυτή η θεματική συγκέντρωση είναι ενόητη και θα πάρουμε αποστάσεις από αυτή την πρόταση. Ε, επενδύσεις λέμε κατά προτεραιότητα και αυτό το 80% δεν έχει νόημα. Τώρα 70, 60, δεν ξέρω, δεν θα παίζουμε την κολοκυθιά τώρα. Υπάρχουν προτεραιότητες, γιατί δεν θα πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Όλοι συνδέονται με τη στρατηγική, ξέρω εγώ, του 2020. Για ποιο λόγο τώρα βάζουμε ποσοστά και δεν ε, θεωρείται προτεραιότητα το ένα ή το άλλο έργο. Ας το αφήσουν αυτό στα επιχειρησιακά σχέδια. Η αστική διάσταση. Μάλιστα. Κανονικά, για να είμαστε σωστοί και καθαροί θα πρέπει να διαγραφεί ο κατάλογος. Συμφωνώ με τον κύριο Σνάιντερ. Και αυτά τα πλατφόρμες και φόρουμ. Υπάρχει Επιτροπή Περιφερειών, συζητάει και τις πόλεις. Ας πούμε να λαμβάνεται περισσότερο η αστική διάσταση υπόψη στην Επιτροπή Περιφερειών και κάτι τέτοια. Νομίζω το καλύτερο είναι να διαγράψουμε αυτό τον κατάλογο. Άρον άρον τώρα βιαζόμαστε να βαφτίζουμε καινούργια πράγματα, να γενιάζουμε καινούργια πράγματα που δεν ξέρουμε γιατί δημογραφική πρόκληση, μάλιστα βεβαίως θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Δεν αρκούν καθόλου αυτά που κάνουν. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις περιφέρειες που έχουν τεράστιο πρόβλημα. Έχουν τεράστιο πρόβλημα και υπάρχουν. Ε, στα ανατολικά σύνορα της Γερμανίας ας πούμε. Θα πρέπει να το σκεφτούμε περισσότερο, ε, όχι να μείνουμε στις προτάσεις όπως έχουν. Ευχαριστώ. Άλλους δύο μιλητές έχουμε σύντομα και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο, Γιάν, και ο Μιχαήλ για να ολοκληρώνω. Κύριε Σφανίστερο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλό είναι που κάνουμε αυτές τις συζητήσεις με συγκεκριμένες τροπολογίες και για το Γενικό Κανονισμό και για το Κανονισμό για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δεν θέλω να επαναλάβω τίποτα. Να ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η εκτίμηση της Επιτροπής Περιφερειών για την ε, υποχρεωτική μεθοδολογία για την ευφυή εξειδίκευση, αυτό το smart specialization. Το έχουν βάλει ως προϋπόθεση. Εσείς τι λέτε γι' αυτό. Το δεύτερο, θα κάνουμε μια ακρόαση το απόγευμα και μια άλλη το Μάιο με ένα θέμα το οποίο δεν έχει εκπονηθεί εγκαίρως ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχει μελετηθεί ε, ορίζον 2020, Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης, Καινοτομία και Έρευνα ε, και η συνέργειά τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει τώρα ένα non-paper για αυτά τα πράγματα. Και ρωτώ, υπάρχουν διαδικασίες εν εξελίξη τώρα στο ορίζον 2020, έχουν βγάλει απ' έξω ε, κάποια κέντρα γνώσης. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υιοθετήσουμε άλλη προσέγγιση. Από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης να έρθουμε και να πούμε ωραία. Αυτό το 80% ας πούμε που δίνουμε για την καινοτομία και τα λοιπά, μας βάζει σε μια άλλη ευρωπαϊκή ατζέντα, την ολοκληρωμένη ατζέντα για τη συνεργασία. Δηλαδή δεν δίνουμε γενικά και αόριστα σε περιφέρειες και πόλεις ε, χρήματα για να κάνουν ευφύ ε, εξυγχρονισμό η εξειδίκευση, αλλά το κάναμε στο παρελθόν στο λεγόμενο στόχο 3, αν θυμάστε, και στο mainstreaming του στόχου 2. Δηλαδή, χρειάζεται μια απάντηση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του καθενός και στραμμένη προς το μέλλον, για να δούμε ε, πώς θα αξιοποιήσουμε το Horizon 2020, τα ε, μέσα για την αριστεία και αυτό που προτείνουμε εμείς. Και σε αυτό το κείμενο δεν βρίσκω τίποτα σχετικό επειδή το συζητάει η Επιτροπή Περιφερειών επανειλημμένα, έχετε εκπονήσει καμία άποψη, έχετε όραμα γι' αυτό και πρόταση, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας στους επόμενους μήνες και καλό είναι να έχουμε όσο γίνεται περισσότερες συμβουλές, να έχουμε και τροπολογίες, θα ήταν ενδιαφέρον κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ένα, ένα μισή λεπτό για Χιμτσέλε. Ευχαριστώ και τον κύριο Σνάιντερ και την Επιτροπή Περιφερειών για την παρατήρηση αυτή, για τα ε, κείμενα της προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμφωνώ. Θα πρέπει να είναι ο κανονισμός ε, ευέλικτος και εφαρμόσιμος και πρακτικός, όχι αυτά τα άκαμπτα που προτείνονται μέχρι τώρα, 5% για τις πόλεις. Συμφωνούμε ότι είναι ειδικό στόχος ενίσχυσης. Ε, μιλήσατε και για περιαστικές περιοχές. Παρακαλώ να συνδεθεί με το πυλώνα 2 της γεωργικής πολιτικής. Δεν χρειάζεται τώρα κάθε χωματόδρομο να τον ασφαλτοστρώσουμε. Ε, και ο πολιτισμός αναφέρθηκε από κάποιους συναδέλφους. Ξέρω ότι θα συμφορήσουν και άλλοι να μπει και ο αθλητισμός ως ε, στόχος ενίσχυσης. Είχαμε την έκθεση για τον αθλητισμό που εγκρίθηκε ήδη από το Κοινοβούλιο και ε, ε, τονίζει και τα διαρθρωτικά ταμεία. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο κοινωνικό ε, και πολιτιστικό κίνημα, αλλά είναι και οικονομική δραστηριότητα και θα πρέπει να ενισχυθεί. παρακαλώ και ελπίζω στην δική σας υποστήριξη και σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Δυόμιση λεπτά, Νικόλας Μάρτιν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο σε αυτή την περίπτωση. Θέλω να επικεντρωθώ σε τρία μεγάλα θέματα. Το θέμα της συγκέντρωσης, το θέμα το αστικό και ε, το δημογραφικό που είναι εγκάρσιο. Για τη συγκέντρωση, ε, σε αυτή την επικεφαλίδα έχουμε εντάξει όχι απλώς ε, τον ειδικό μηχανισμό για τη θεματική συγκέντρωση αλλά και τις μεγάλες επιχειρήσεις και τη βασική υποδομή. Τι λέμε εδώ και πού βασίζεται η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τη χρήση των κονδυλίων. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να κάνουν επιλογέ. Πώ θα χρησιμοποιούν τα κονδύλια. Δεν θα πρέπει οι πάντε να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τα πάντα, αλλά να δουν πώ θα πιάσουν τόπο τα κονδύλια για να επιτευχθούν οι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό έρχεται να δικαιολογήσει για την, την εξαίρεση της χρηματοδότησης για ε, παραγωγικές επενδύσεις των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξαιρούνται από παντού. Ε, στην έρευνα, στην τεχνολογία μπορούν να ενταχθούν. Αλλά παραγωγικές επενδύσεις ε, περιορίζονται αυτές στις μικρομεσαίες, κυρίως για την Υποδομή επίσης, βασική υποδομή στις πιο αναπτυγμένες ε, περιοχές δεν μπορούν να πηγαίνουν κοινοτικά κονδύλια γιατί υπάρχουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης. Ο μηχανισμός του άρθρου 4 είναι εκ των όνου κάνευτο. Ε, αναφέρει συχνά ο Επίτροπος Χάν ε, στην εστίαση και στην ευελιξία. Χρειαζόμαστε εστίαση και ένα μηχανισμό για να επιτευχθεί αυτή και θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι στοιχειώδεις περιορισμοί στον κανονισμό. Δεν μπορεί να είναι μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω ε, με αναδιαπραγμάτευση κάθε φορά. Δεν λειτουργεί αυτό. Βεβαίω θέλουμε να υπάρξει μια ευελιξία, αλλά ε, με συγκεκριμένη εστίαση και στόχευση. Ε, κάθε φορά να κοιτάμε αν χρειάζεται, αν είναι δικαιολογημένη κάποια επέκταση. Για το θέμα των πόλεων, όπως σας είπα χτες, γονέκυψαν και συζητήθηκαν τα ίδια θέματα στην Επιτροπή σας, σε άλλη έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη να ξανακοιτάξει αυτό το θέμα του καταλόγου πόλεων, να μιλήσουμε για αρχές και μεθοδολογία. Για την πλατφόρμα της αστικής ανάπτυξης νομίζω ότι αιτιολογείται, διότι θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο των όσων προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 5% ως κατόφλι για ολοκληρωμένες δράσεις για η φόρο ανάπτυξη των πόλεων που συνδέεται και με τις καινοτόμε δράσεις σε αστικές περιοχές. Η πλατφόρμα θα μπορούσε να είναι ένα τρόπο συνεργασία όλων των πόλεων που έχουν υιοθετήσει αυτές τις δράσεις για να προωθηθεί και να ενθαρρυνθεί η επιτυχία. Εμείς δεν θέλουμε καμία αποκλειστικότητα στην πλατφόρμα, να συμμετέχουν όλες οι πόλεις που έχουν αυτές τις δράσεις. Και ένα τελευταίο για τη δημογραφική πρόκληση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό είναι ένα θέμα εγκάρσιο και αφορά διάφορες πολιτικές και θα πρέπει να ε, το δούμε στην ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις εδαφικές ανάγκες που έχουν εγγραφεί σε όλη ε, τη στρατηγική και τον προγραμματισμό. Και έτσι δρομολογούνται και οι επιλογές για τη χρηματοδότηση για ειδικές θεματικές ε, ενότητες και επενδυτικές προτεραιότητες. Ευχαριστώ. Ο Μίχαελ Σνάιντερ. Äh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να τονίσω ότι ε, ε, έχω εντυπωσιαστεί από την ευρεία συνένεση που επετεύχθη και είναι πολύ ευχάριστο όταν άτομα τόσων διαφορετικών περιφερειακών προελεύσεων και πολιτικών προελεύσεων ε, συνενούν δείχνει το ύψος της αξιοπιστίας και ε, βεβαίως θέλω να τονίσω ότι βεβαίως οι περιοχές που είναι κοντά στην πόλη και κοντά στην Ήπερθρο θα πρέπει να συνυπολογιστούν στον προγραμματισμό. Δηλαδή η πόλη δεν μπορεί να ε, εξεταστεί μονοπλευρά και απομονωμένα. Επίσης ε, το σημειώνω την υπόδειξη για την γνωμοδότησή μου και θα κάνω μια σχετική τροπολογία στην Ολομέλειά μας και θα θίξω το θέμα αυτό. Ε, επίσης, δημοκρατική πρόκληση. Ό,τι και να πούμε, οι δημοκρατικές περιφέρειες θα χρειαστούν και στο μέλλον βοήθεια και αυτό αναφέρεται άλλωστε και στη συνθήκη της Λισαβόνας. Διαπιστώνουμε όμως ότι υπάρχουν και νέες μορφές δημογραφικών προκλήσεων που περιλαμβάνονται τώρα στην περιφέρεια αλλά ίσως σε 10 χρόνια δεν θα είναι πλέον περιφερειακές ε, κατόπιν των αλλαγών των δημογραφικών. Άρα ε, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την ευελιξία κατά τρόπον ώστε να απαντήσουμε επικοδομητικά στις περιφέρειες ε, και γι' αυτό βλέπουμε σαν παράδειγμα γιατί ο θεματικός περιορισμός δεν ε, μπορεί να ανταποκριθεί ή στις ε, επιταγές της εκάστοτε καταστάσεως. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι θέλετε κάτι να πείτε, αλλά ευχαρίστω αν θέλετε. Νομίζω ότι υπάρχει μόνο ένα θέμα που έχει μείνει ακόμη σε κρεμότητα, η πλατφόρμα των πόλεων και πιστεύουμε ότι χρειάζεται μία παρακολούθηση της δράσης. Το ερώτημα είναι χρειαζόμαστε να δημιουργήσουμε μέσω νομοθετικού κειμένου ένα νέο όργανο διότι ουσιαστικά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συζητήσουμε και το πρόβλημα για τις ε, επιχειρήσεις. Ναι, ας ελπίσουμε ότι θα λεχθεί ότι δεν θα μειώσουμε κατά αυτόν τον τρόπο την εξέλιξη των πόλεων και έτσι κλείνω το θέμα αυτό, φτάνουμε στο 17 του κυρίου Μπουστινάρου αλλά θα ξεκινήσουμε με τον Ρωμαίου Σταβαράτσε που είναι εδώ, δηλαδή την παρουσίαση της Επιτροπής Περιφερειών και θα έχουμε περιορισμένο χρώμα τον οποίο σας αναφέρω. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι με καλέσατε εδώ να συμμετάσχω στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ιδιαίτερη τιμή ότι εκπροσωπώ το, την Επιτροπή Περιφερειών για το νέο, το νέο θέμα ε, όσον αφορά την διαδικασία ε, εφαρμογής και ε, και βελτίωση ε, ομίλων διότι βλέπουμε ότι εδώ αντικατοπτρίζονται οι απόψεις των περιφερειών διότι το Ταμείο Συνοχής αποτελεί για όλους μας ε, ένα βασικό θέμα ε, και με τα μέσα αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν τα μεγάλα περιβαντολογικά προγράμματα υποδομής και και ιδίως στις λιγότερες ανεπτυγμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Χωρίς αυτή την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αυτά τα προγράμματα δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Δεν χρειάζεται εδώ να αναφερθώ εις ε, την σημασία για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να περιλάβω και την προσωπική μου άποψη ότι για να μπορέσουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί θα πρέπει να δώσουμε σε όλες τις περιφέρειες ίδιες δυνατότητες ε, είτε, είτε πρόκειται για πιο ανεπτυγμένες είτε για διαρθρωτικά πιο ασθενείς θα πρέπει να διευκολυνθούν να υλοποιήσουν όλες τους τις δυνατότητες και γι' αυτό στην ε, ε, γνωμοδότησή μου αναφέρω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι προτεραιότητες είναι σημαντικές για να μπορέσουν να συνδέσουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για καλύτερη λειτουργία της Ευρώπης και για ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και για την αλληλεγγύη με τις διαρθρωτικά πιο ασθενείς περιοχές. Θέλω εδώ να τονίσω ένα βασικό θέμα και ελπίζω να με στηρίξετε. Είναι η υποχρεωτική εμπλοκή όλων των κυβερνήσεων και διοικήσεων σε ένα τέτοιο ισοσκελισμένο ε, κοινωνικό επίπεδο με τη βοήθεια της επικουρικότητος αλλά οι πόλεις δεν, θα δεν συμμετέχουν επαρκώς στη λήψη των αποφάσεων όχι τουλάχιστον όταν πρόκειται για μεγάλα προγράμματα μεταφορών τα οποία χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρομαι εδώ στα TNT, στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Χρειαζόμαστε λοιπόν νέες αρμοδιότητες Χρειαζόμαστε ένα νέο πλαίσιο για να μπορέσει να υπάρξει εδαφική συνοχή και για να μπορέσουν να προωθηθούν και οι δευτερεύουσες διασυνδέσεις και ευρωπαϊκά και περιφερειακά. Πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι και στην γνωμοδότηση μου προτείνω οι επενδύσεις στα ενεργειακά ε, οικονομικά ε, κτίρια να χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλο που ένα μέρος χρηματοδοτείται από το ΕΦΡ δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά περιοριστικοί διότι υπάρχουν θέματα που έχουν τοπικό ή περιφερειακό ενδιαφέρον και θα πρέπει ε, να ε, μην ξεχνούμε ότι υπάρχει μία πληρέστερη εικόνα από, την οποία, από αυτή που έχουμε ίσως από μακριά. Επίσης όσον αφορά τη βιωσιμότητα ορισμένων επενδύσεων. Ναι μεν στηρίζουμε ε, τον φιλόδοξο στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία, ε, ε, το οποίο έχει καταγράψει στο χάρτη πορείας των μεταφορών να μειώσει τις εκπομπές κατά 60% αλλά θα πρέπει όλα αυτά να έχουν συνδυαστεί και εξεταστεί από όλες τις πτυχές μακροπρόθεσμα. Όσον αφορά την βιωσιμότητα των ε, επενδύσεων και τις περιβαλλοντολογικές απόψεις, όπως σας είπα, στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρομαι εδώ στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές, όπου μιλάμε ότι ε, για τη μείωση των ε, εκπομπών κατά 60% ως το 2020 και ε, αυτό να ε, γίνει με ε, πόρους του Ταμείου Συνοχής. Πρέπει όμως να αξιολογηθεί η μακροπρόθεσμη απόδοσή τους και θέλω τώρα να αναφερθώ εις το μέσο δικτύωσης της Ευρώπης που αποτελεί μια καινοτομία πρόκειται για μια ένα νέο κίνητρο για τον προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση διασυνοριακών προγραμμάτων μεταφορών ενεργείας ε, και ε, ε, πρόκειται για 10 δισεκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων το 20% προέρχεται από το Ταμείο Συνοχής.

Ε, το, ο κανονισμός για αυτό το μέσον προβλέπει ότι θα χρησιμοποιηθούν ε, στις σιδηροτροχές ε, στα κράτη-μέλη βάσει της νομοθεσίας η οποία υπάρχει σε εθνικό επίπεδο πράγμα το οποίο συνάδει με τους στόχους της στρατηγικής για το 2020 όπου θέλουμε να ολοκληρώσουμε ολοκληρώσουμε, ολοκληρώσουμε τα προγράμματα για την εσωτερική αγορά ε, και πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διασύνδεση μεταξύ των περιοχών. Θεωρούμε όμως ότι το μέσο αυτό ναι μεν έχει μία σημαντική προστιθέμενη αξία, δημιουργεί θέσεις εργασίας, αλλά ε, πέραν αυτής της πρωτοβουλίας η οποία ε, καταγράφεται στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμπεριλάβει ε, και ιδιωτικά κεφάλαια. Δηλαδή ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελήσει το κίνητρο για να συμπαρασύρει τις ε, ιδιωτικές επενδύσεις κατά την ε, προετοιμασία και κατάρτιση ορίμων προγραμμάτων ε, θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη σωστής διαχείρισης και εδώ έχουμε ορισμένες ε, επιφυλάξεις εις την Επιτροπή Περιφερειών ιδίως όσον αφορά τη χρήση των 4 δισεκατομμυρίων από το, το Ταμείο Συνοχής διότι εξυπηρετείται κάτι το οποίο δεν προωθεί προωθεί την ε, ε, συνεργασία και την ε, ε, το συντονισμό των προσπαθειών ε, ενώ πιστεύουμε ότι θα έπρεπε τα 10 δισεκατομμύρια ε, να δοθούν στις πόλεις μέσω των αρμοδίων οργανισμών ενώ ο Επίτροπος Κάλλας μας είπε ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ευρωπαϊκά. Τώρα εσείς θα αποφασίσετε και εμείς πρέπει να εποπτεύουμε τα προγράμματα να εφαρμοστούν σωστά, να ε, κινητοποιηθούν και να μπορέσουμε να επιτύχουμε διότι διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος η δυνατότητα αυτή να μην συμβάλλει εις ε, την ε, διασυνοριακή συνεργασία. Η Επιτροπή Περιφερειών είναι υπέρ μιας πολιτικής συνοχής η οποία θα είναι ισχυρή και ε, χρειάζεται και μία σωστή πολιτική συνοχή, γι' αυτό και παρακαλούμε ε, να μην μειωθούν οι πόροι για το Ταμείο Συνοχής στον επόμενο προϋπολογισμό πράγμα το οποίο θα ήταν μία επιστοδρόμηση σε σχέση με το παρελθόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Πίκτορ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως καλωσορίζω όσα είπε ο κύριος Σταβαράκη, ε, δήμαρχος του Βαρό, από τη Ρουμανία. Νομίζω ότι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί και οφείλει να στηρίξει αυτή τη φιλοσοφία γιατί είναι η μόνη που μπορεί να στέψει με επιτυχία την επόμενη προγραμματική περίοδο. Τα σχόλια ε, στην έκθεσή μου ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τα σχόλια του κυρίου Σταβαράκη. Θα ασχοληθώ όμως σε μερικά στοιχεία επί των οποίων θέλουμε ε, αμοιβαία στήριξη και τα σημεία επί των οποίων ενωμένη η Επιτροπή μας με την Επιτροπή Περιφερειών θα πρέπει να πείσει το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Ένα στοιχείο σχετικά με, την, ε, ε, με το μέσο Connecting Europe. Αμφιλεγόμενο και πολύ συζητημένο. Εγώ ως εισηγητής είμαι υπέρ αυτού του προγράμματος. Είμαι υπέρ της οικοδόμησης μιας τέτοιας φιλοσοφίας που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε προβλήματα ε, που αφορούν διασυνοριακά ζητήματα. Είμαι υπέρ της μεταφοράς των 10 δις από το Ταμείο Συνοχής στο μέσο Connecting Europe. Αλλά υπάρχει ένα όμως. Ένα όμως το οποίο δεν είναι κατά του προγράμματος, όμως αφορά την έλλειψη εγγυήσεων που χρειάζομαστε και εμείς ως βουλευτές και το, και η Επιτροπή Περιφερειών. Βεβαίως πρέπει να ξεκινήσουμε διάλογο με την DG Move που διαχειρίζεται το μέσο Connecting Europe. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις και στο Συμβούλιο. Το ίδιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τολμώ να πω. Υπάρχουν επίσης και διστάμινες απόψεις και στην Επιτροπή μας εδώ. Ο μόνος τρόπος για να σώσουμε τη φιλοσοφία του μέσου Connecting Europe, ε, το μόνος τρόπος για να σώσουμε λοιπόν το πρόγραμμα αυτό είναι να γεφυρώσουμε την ε, ε, φιλοσοφία της συνοχής με την φιλοσοφία της Digimove που αυτή επιβάλλεται αυτή τη στιγμή. Να καθίσουμε μαζί όλοι και να προσπαθήσουμε να βρούμε μία έκβαση ε, καλύτερη. United and we shall solve και με τους συναδέλφους της Επιτροπής ε, Μεταφορών έτσι ώστε να ε, ξεπεραστούν τα ερωτήματα τα οποία παραμένουν αναπάντητα καθώς επίσης και κάποιες ζώνες έτσι σκιάς και αμφιβολίας ε, γιατί μόλις λυθούν τα προβλήματα αυτά τότε είμαστε σαφώς υπέρ. Επίσης όσον αφορά την στήριξη της ενεργειακής απόδοσης. Συμφωνώ απολύτως, μπορώ να προσθέσω μόνο ότι κατά την άποψή μου αυτό είναι ουσιώδες. Θα πρέπει να επιτύχουμε τους στόχους του 2020 και υπάρχουν άλλωστε πολλές μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης των εκπομπών και ορθής χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Βεβαίως γνωρίζω ότι υπάρχει στήριξη για το θέμα αυτό. Στο Συμβούλιο υπάρχει και ευελιξία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, κάνω έκκληση και σε εσά μαζί με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, την Επιτροπή Ρέτζη, να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση έτσι ώστε να υπάρξει πρόσβαση στο Ταμείο Συνοχής για θέματα ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης. Ε, τρίτον, να δώσουμε δυνατότητα χρήσης των χρημάτων του Ταμείου Συνοχής ε, για την οικοδόμηση ε, εγκαταστάσεων για την παραγωγή ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί στα νοικοκυριά. Ε, επίσης ε, να μειωθούν, με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν και τα, ε, τα αέρια του θερμοκηπίου και βεβαίως θα δοθεί και όθηση όσον αφορά τη βελτίωση του ενεργειακού μείγματος που θα επιτρέψει τελικά την μείωση των λογαριασμών ενέργειας που σε όλες τις χώρες αλλά κυρίως στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη αρχίζουν να γίνονται ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ένα επόμενο σημείο, και εδώ κάνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να διασφαλίσει ότι θα έχουμε λύσεις έτσι ώστε να αυξηθούν οι διοικητικέ ε, ε, δυνατότητες, ε, ικανότητε. Χθε συζητήσαμε το θέμα αυτό. Είναι τόσο περίπλοκα τα θέματα αυτά. Νέοι οργανισμοί θα ιδρυθούν και θα αρχίσουν να λειτουργούν το 2013. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί θα λειτουργούν καλά και αποτελεσματικά και πλήρως τον Ιανουάριο του 2014. Εάν δεν έχουμε όμως διασφαλίσεις ότι η ικανότητα διοικητική και θεσμική θα αυξηθεί, τότε, τότε θα έχουμε τον ίδιο κατάλογο που, είχαμε, που πήραμε σήμερα όπου πάρα πολλές χώρες έχουν ε, σταματήσει τις διαδικασίες. Το βλέπουμε αυτό, το γράφει δίπλα στα ονόματά του στον κατάλογο. Ε, πρέπει να βελτιώσουμε λοιπόν τις ικανότητες έτσι ώστε να επιτύχουμε τα σχέδιά μας αυτά. Ε, διάλογος επίσης με, με όλα τα σώματα σε τοπικό εθνικό επίπεδο. Ε, και οπωσδήποτε σαν απόρριο των συζητήσεων αυτών έχουμε την καλύτερη πρόσβαση των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες ε, σε όλες τις ε, διεργασίες. Θα πρέπει να το δούμε γιατί λείπει, λείπει αυτή η αναφορά στην πρόταση κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής και θα ευθυγραμμιστούμε με τον τρόπο αυτό και με, την, με το μέσο Connecting Europe καθώς επίσης και με όλους τους άλλους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Τέλος, Λυπούμε γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή ο Επίτροπος Ποτόσνικ δεν κατάφερε να ε, παρουσιάσει δημόσια την, ε, τη νέα έκδοχη ε, και την μελέτη αξιόλογης, στρατηγικής αξιολόγησης και επίπτωσης. Είχαμε μια παρόμοια συζήτηση και με την Επιτρόπο Χέντεγκάρτ πιστεύω ότι θα πρέπει να ελεγχθεί και να εφαρμοστεί κανονικά βεβαίω το κανονιστικό πλαίσιο μετά το 2014, αλλά θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ταυτόχρονα ότι ευθυγραμμίζονται όλες οι προσπάθειές μας με το περιβάλλον, με την κλιματική αλλαγή και με την βιοπικιλότητα, γιατί διαφορετικά ε, θα είναι δύσκολο μέσα σε αυτούς τους, νέου νέους κανόνες ε, να ε, απομονώσουμε όλα τα στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν καλό τον Επίτροπο να το κάνουμε τώρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε στους κανόνες μας αυτές, αυτούς τους νέους κανονισμούς και αυτές τις νέες ιδέες, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι η φιλοσοφία μας θα είναι διαρκής, συνεχής και συνεκτική. Αυτά ήθελα να σας πω, οι απόψεις της Επιτροπής βεβαίως ε, θα μου είναι πολύτιμες και βεβαίως να εκφράσω για μία ακόμα φορά την ευγνωμοσύνη μου προς την Επιτροπή των Περιφερειών για την σαφή και διαρκή του δέσμευση. Συνάδελφοι, δέκα λεπτά έχουμε για τη συζήτηση, ξέρετε. Αν έχετε τίποτα γρήγορε ερωτήσει για την Επιτροπή Περιφερειών, γιατί μετά τι 5 την ακρόαση δηλαδή θα συνεχίσουμε, αλλά θα απουσιάζει η Επιτροπή Περιφερειών. Η κυρία Κλάουδια Σμιτ ε, έχει ε, φτάσει ήδη η Ομοσπονδιακή Υπουργό Παιδεία, Τεχνών και Πολιτισμού τη Αυστρία και στι 12 προβλέπεται συζήτηση μαζί τη. 10 λεπτά παρακαλώ έχουμε. Αν έχετε να πείτε τίποτα για την Επιτροπή Περιφερειών σα παρακαλώ. Ε, τα υπόλοιπα θα τα δούμε με τον Βίκτορα το βράδυ. Η κυρία Ματσόνη και ο Λάμπερ Φανίστερο είναι τη σειρά αυτή ή αντίστροφα όπως θέλετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αρμόδια επιτροπή της Επιτροπής Περιφερειών μας παρουσίασε σήμερα μια εξαιρετική ε, εργασία και φαντάζομαι ότι και στην Ολομέλεια ε, θα υποβληθούν τα ίδια στοιχεία τα οποία ευθυγραμμίζονται βεβαίως με τις δικές μας ευαισθησίες και τις δικές μας ανησυχίες. Μας ε, ικανοποιεί λοιπόν αυτή η ταύτιση απόψεων. Θα ήθελα να πω δύο λόγια σχετικά με το σημείο σχετικά με, τις, με την αιρεσιμότητα. Αυτό αναφέρεται και στην γνωμοδότηση την οποία μελετούμε και θα ήθελα ιδιαίτερα να ζητήσω από τον Πρόεδρο σε αυτήν την μακροοικονομική αιρεσιμότητα και, την διασύν... και τη... σε σχέση με την διασύνδεσή τους με τις παραμέτρους ε, του Μάστριχτ, ε, την πολιτική συνοχή και τους κανόνες διακυβέρνησης εν να μου πούν ποια είναι η άποψή τους, ε, ξεκινώντας βεβαίως από το γεγονός ότι το Ταμείο Συνοχής έχει ήδη επιβαρυνθεί με αυτές τις στρατηγικές προβλέψεις και ότι από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζουμε βεβαίως και ειδικέ περιπτώσεις όπως ας πούμε την Ουγγαρία, χώρα για την την οποία πρώτη φορά εφαρμόστηκε η άρση των, ε, των χρημάτων του Ταμείου γιατί ε, ξεπέρασε το 3% που προβλέπεται από τη συνθήκη του Μάστριχτ. Δεύτερο σημείο. Σχετικά με το ΣΕΦ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε με την ανησυχία που εξέφρασε ήδη η Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τον ασαφή τρόπο ε, που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για διαχείριση αυτών των πόρων κυρίως δε όσον αφορά τον τελικό στόχο αυτών των ταμείων, αυτών των πόρων, συγγνώμη, ε, που λαμβάνονται από τις διάφορες χώρες, δηλαδή που θα ήταν θεωρητικά στη διάθεση κάποιων χωρών και που δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο ακριβώς θα ανακατεμηθούν. Εάν θα χρησιμοποιηθούν δηλαδή τελικά στην χώρα προέλευσης ή και σε άλλες χώρες. Και εδώ επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το βλέπω αυτό να υπογραμμίσουμε και δεν το βλέπω να υπογραμμίζεται ιδιαίτερα στην Επιτροπή Περιφερειών και στο έγγραφό τη, Να υπογραμμίσουμε, λέω, την ε, ανάγκη πιο ακριβούς ε, ε, πρόβλεψης της χρήσης των κονδυλίων από άλλα ταμεία όταν αναφερόμαστε στις ίδιες, ε, ε, στα, στα ίδια προγράμματα, δηλαδή προστασία περιβάλλοντος και δημιουργία υποδομών. Ευχαριστώ πολύ, Λέμπερ Βανίστερόι. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίως για την ομόφωνη τοποθέτηση της έκθεσης της Επιτροπής Περιφερειών. Καλό είναι να συνεχίσουμε και αυτά που ορίζονται στη συνθήκη. Ιδιαίτερη προσοχή στα νέα κράτη-μέλη ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, το περιβάλλον και τις μεταφορές. Δύο σημαντικά ζητήματα. Την περασμένη φορά είχα πει κάτι, την πρώτη φορά που συζητήσαμε αυτό το θέμα, για το εξή γεγονός. Καλή η υπόθεση των υποδομών, αλλά αν κοιτάξουμε σε 10, 20 και 30 χρόνια, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι οι φυσικές υποδομές, αλλά οι υποδομές της γνώσης που θα πρέπει να προωθούν αυτές οι χώρες και να τις προαγάγουν. Και εκεί η ανταγωνιστικότητα και ο ανταγωνισμός είναι ο ίδιος με τα παλιά κρατημέλη. Γιατί λοιπόν στις μεταφορές και στις υποδομές δεν το επεκτείνουμε στις υποδομές της γνώσης. Τα παλιά κρατημέλη έχουν 90% των κονδυλίων της έρευνας και της ανάπτυξης και παραμένει αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να δεχθούμε από πλευρά συνταφικής συνοχής, να μην πηγαίνουν αυτά τα χρήματα ε, στις νέες χώρες. Καλό το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία για την ενεργειακή απόδοση, την έρευνα στις υποδομές, στις ε, φυσικές πραγματικά σκληρές υποδομές, αλλά και στις υποδομές γνώσης. Αυτό θα προωθήσει και θα αναπτύξει περισσότερο αυτές τις χώρες. Ξέρω ότι είναι δύσκολο νομικά να κατοχυρωθεί κάτι τέτοιο σε ένα κείμενο, αλλά και είναι τα χοντρά λεφτά για να το πω έτσι. Γιατί έχουμε την παλιά νοοτροπία και δεν αντιμετωπίζουμε τις νέες προκλήσεις ε, και η Επιτροπή Περιφερειών. Και ο εισηγητής μου πώς θα μπορούσε να μας απαντήσει, γιατί αυτό με απασχολεί. Could, could you please, I mean, Σας ευχαριστώ. Δεν Εάν ε, η Κορνέλια θέλει να πει κάτι, αλλά θα ήθελα να πω για μία ακόμα φορά επικεντρωθείτε τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή Περιφερειών. Ναι, ο κύριος ε, Χρυσόγελος, ε, θα πω δύο λόγια τώρα σε σχέση με την Επιτροπή Περιφερειών. Θα ήθελα να θίξω και τα υπόλοιπε ερωτήσει μετά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, όχι να μιλάμε γενικά για υποδομές, ε, αλλά για ε, αηφόρο, αϊφόρο συγγνώμη, υποδομές σε σχέση με άλλες διαδοτικές πολιτικές. Νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό το σημείο. Εάν συζητήσουμε για μεταφορές, ας πούμε, θα πρέπει να αναπτύξουμε ιδέες και προγράμματα για αηφόρο μεταφορά. Επίσης, αν μιλάμε για ενέργεια, θα πρέπει να είναι ε, αηφόρος ε, ε, ενέργεια, ανανεώσιμη ας πούμε. Όχι γενικόλογα λοιπόν, θα ήθελα περισσότερη αστίαση για το θέμα αυτό. Κορνέλη, θες να προωθήσεις κάτι? It's okay. So, discuss we can later on, but... Εντάξει, θα το συζητήσουμε μετά. Πολύ σύντομα, μία, μία μόνο ερώτηση. Αυτό το μέσο Connecting Europe, δεν έχω καταλάβει ακριβώς η Επιτροπή Περιφερειών τι άποψη έχει. Γιατί είναι κεντρική η διοίκηση. Τελείως διαφορετικό το σύστημα που σχεδιάζεται με ΑΙ τώρα. Η Επιτροπή Περιφερειών ε, τι άποψη έχει γι' αυτό και σε σχέση με το Ταμείο Συνοχής. Ευχαριστώ. Ο κύριε Σταβαράτσα, αν θέλετε να απαντήσετε, παρακαλώ. Γιατί σας έγινε ερώτηση για τη μακροοικονομική αρισιμότητα. <clears throat> Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να σας πω ότι η θέση της Επιτροπής των Περιφερειών είναι προς την ίδια κατεύθυνση με τα όσα είπε εδώ ο κύριος Μποστινάρου. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με την πρόταση αυτή. Πολύ καλή ιδέα οι επενδύσεις να ε, ε, πηγαίνουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί είναι μια καλή αφετηρία. Συμφωνούμε λοιπόν απολύτως με αυτά που προτάθηκαν. Κάτι άλλο που θα ήταν σημαντικό πέρα από αυτά είναι να δούμε και ποιες είναι οι διοικητικέ δυνατότητες στα πλαίσια μιας τέτοιας ανάπτυξης. Δηλαδή, οι ε, αρχές που καλούνται να διχειριστούν αυτά τα πράγματα θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν τη σωστή κρίση, να παίρνουν σωστές αποφάσεις ε, για να βελτιώνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός. Ότι υπάρχει δυνατότητα στη διοικητική μηχανή, σε επίπεδο τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, να διαχειριστούν αυτά τα προγράμματα και οι πραγματικοί δικαιούχοι να υποφελούνται. Ειδικά λοιπόν η τεχνική βοήθεια θα πρέπει να συντονιστεί καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, ανέκαθεν αποδεικνύεται αυτό ότι κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε. Δεν θα πρέπει να κατακαιρματιστεί η τεχνική βοήθεια. Ε, διαπιστώθηκε και αποδείχτηκε μάλιστα ότι το πρόβλημα εστιάζεται εκεί σε πολλά κράτη-μέλη. Για την ερώτηση κυρίας Ματσόνη τώρα. Η χρήση άλλων πόρων. Κοιτάξτε, δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς εκεί είμαστε πρόθυμοι να το συζητήσουμε. Και να συμπεριλάβουμε τις σκέψεις αυτές στην έκθεσή μας. Για την μακροοικονομική αιρεσιμότητα, δηλαδή να υπάρχουν κάποιοι όροι και προϋποθέσεις ε, στα κονδύλια, ξέρουμε ότι όταν έχουμε τέτοιες απαιτήσει και προϋποθέσεις. Μπορεί να γίνει αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν μπορεί η πολιτική συνοχή να είναι ένα μέτρο διόρθωση των σφαλμάτων των κρατικών προϋπολογισμών. Υπάρχουν κάποιοι στόχοι, υπάρχουν κάποιε προτεραιότητες, τα αντίστοιχα άρθρα και μάλιστα τη συνθήκη της Σαββόνας για το τι είναι η συνοχή, ε, άρθρο 171, 174 και επόμενα. Θεωρούμε λοιπόν ότι η μακροοικονομική αιρεσιμότητα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και υποχρεωτικά για όλα τα κεφάλαια όμως του προπολογισμού, όχι μόνο για εκείνα που αφορούν τη Ταμείο συνοχή. Όλοι να έχουμε την ίδια θέση, αυτό θα μπορούσε τότε και μόνο τότε να αποτελέσει μια καλή αφετηρία για τη συζήτηση. Δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να τιμωρείται ένας τομέας και να είναι συνοχή και ιδιαίτερα η Δήμη, εν αυτά τα μακροοικονομικά είναι τελικά κρατική ευθύνη και όχι τη τοπική αυτοδιοίκησης. Για τον κύριο Φανίστελ Ρόι. Εμείς υποστηρίζουμε την αρχή και τη σκέψη που λέει ότι θα πρέπει να επενδύουμε και στην υποδομή της γνώσης. Όχι μόνο στην ενεργειακή απόδοση και στις φυσικές υλικές υποδομές. Συμφωνούμε με τον κύριο Βανιστερόη ότι θα πρέπει να επενδύουμε και στις υποδομές της γνώσης, αλλά δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα βλέπει κανείς σε ένα γενικό πλαίσιο, σε ένα συνολικό πλαίσιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα είναι να καλυφθούν οι ανάγκες των περιφερειών και των δήμων και κοινοτήτων. Αλλιώς θα έχουμε χάσει το στόχο μας. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε την Επιτροπή Περιφερειών που μοιράστηκε μαζί μας τις σκέψεις αυτές για τα Ταμεία Συνοχής. Αν χρειάζεται, μετά τις 5 θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Αλλά τώρα θα ήθελα να καλέσω στο Προεδρείο την Υπουργό και στο μεταξύ θυμίζω στους συναδέλφους ότι πριν από λίγο καιρό ε, είχε προτείνει η Κωνσταντσε Κρέλ το εξής. Για πρώτη φορά στην ιστορία ε, της συνοχής η αυστριακή κυβέρνηση ε, έκανε μια έκθεση για το ρόλο τεχνών πολιτισμού σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο. Η κυρία Σμίτ είναι η Ομοσπονδιακή Υπουργό Παιδεία Τεχνών και Πολιτισμού και θα ήθελα να μα παρουσιάσει αυτέ τι προτάσει για το τι έγινε στην Αυστρία, πώ πήγε η κατάσταση αυτή και εμεί τώρα που εκπονούμε ε, τις μελλοντικές προστάσεις ε, με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να μάθουμε από την Αυστρία ε, όλα αυτά τα επιτεύγματά της. Καλώς ορίσατε και έχετε μέσα στο λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σήμερα να ε, σας μιλήσω διότι αναφέρομαι στον ρόλο της ε, τέχνης και του πολιτισμού στον τομέα της ε, περιφερειακής πολιτικής διότι ε, η ε, τέχνη και ε, ο πολιτισμός δίνουν την ιδιομορφία των περιοχών και συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής, στην ευημερία και στην ευχάριστη διάθεση των πολιτών της Ευρώπης. Πράγμα το οποίο μπορούμε να επιτύχουμε μόνο εάν ε, ε, κάνουμε μία συζήτηση επί των πνευματικών αξιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ο τομέας του πολιτισμού και των τεχνών κατά τη γνώμη μου και θα επανέλθω στην μελέτη σε λεπτομέρειες ε, δεν πρέπει να περιορίσουν τις ε, δυνατότητές τους θα πρέπει να προωθήσουν την ανάπτυξη, την καινοτομία, να βελτιώσουν το κάλος των ε, περιοχών και να συμβάλλουν στην συνοχή. Και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν, ε, μπορεί ο πολιτισμός, ε, το θέμα του πολιτισμού να συμβάλλει ή στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής του 2020 και όσον αφορά την ε, μελλοντική μας πολιτική το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει μία νέα έννοια για την καινοτομία που δεν ε, θα περιορίζεται μόνο στην τεχνολογική καινοτομία αλλά θα αφήσει πολύ χώρο ε, για τις δυνατότητες της δημιουργικότητας της τέχνης και του πολιτισμού στο βιομηχανικό σχέδιο σχέδιο ή στην αρχιτεκτονική μέχρι και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οπότε με αυτόν τον τομέα και σε αυτόν τον τομέα θα υπάρχει μία έξυπνη εξειδίκευση ε, των περιοχών και η τέχνη και ο πολιτισμός όπως άλλωστε και η δημιουργική οικονομία μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας. Οι διαπραγματεύσεις για την νέα περίοδο προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως βρίσκονται τώρα σε μία αποφασιστική στιγμή. Υπάρχουν νέα θέματα τα οποία τίθενται και υπάρχουν πολύ καλά ε, επιχειρήματα για να μπορέσει κανείς να εμπλέξει περισσότερο κανείς τα πολιτιστικά θέματα στην περιφερειακή ανάπτυξη. Γι' αυτό και στη χώρα μου ζητήθηκε να κάνουμε μία μελέτη από το Υπουργείο μας για ε, ε, τα δημιουργικά προγράμματα και ε, για την συμβολή του στην ανάπτυξη της Αυστρίας. Ε, το Νοέμβριο του 2011 από κοινού με τον Επίτροπο Χάν παρουσιάσαμε στη Βιέννη αυτή τη ε, μελέτη, τη συζητήσαμε, ήταν ενδιαφέρουσα και ήταν συγχρόνως μια πολύ ενθαρρυντική συζήτηση και είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσω και προς εσάς που είσαστε νομοθέτης να σας μεταφέρω τα πέντε βασικό σημεία της μελέτης αυτής από τη δικιά μου σκοπιά. Και πρώτον, ο πολιτισμός ε, μπορεί ε, να συνδυαθεί σε πολλά θέματα ή στην Αυστρία. Δεύτερο θέμα, στον χρόνο της μελέτης, δηλαδή 2007 έως 2010, διαπιστώσαμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον πολιτισμό στην Αυστρία ε, είχαν ε, αποδοθεί 79 εκατομμύρια ε, ευρώ για να επενδυθούν σε πολιτιστικά προγράμματα ή στην Αυστρία και αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό για τη χώρα μου είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Θα ήθελα εδώ να τονίσω το, την δυνατότητα για μικρά προγράμματα που μπορούν να στηρίξουν πολιτιστικές εκδηλώσεις και να αυξήσουν το, ε, ε, ε, την ομορφιά των περιοχών. Επίσης δίνεται μία σημαντική όθηση στην απασχόληση στην Ευρώπη και έτσι και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αντιμετωπίζει όλο και περισσότερες αιτήσει. και με αυτήν τη δημιουργική οικονομία μπορούν να προωθηθούν και ε, οι ε, θέσεις των ε, συνεργατών στα εγχειρήματα αυτά και επίσης το πέμπτο θέμα είναι οι δημιουργικοί πόροι οι οποίοι μπορούν να εξοικονομηθούν από παραδοσιακές πηγές και να χρησιμοποιηθούν ε, σε, νέες, ε, σε νέους τομείς όπως τους συνεταιριστικούς πολιτιστικούς τομείς παραδείγματος χάρη. Θα αναφέρω εδώ τρία παραδείγματα στα πλαίσια της, του Ταμείου Συνοχής που συγχρηματοδοτήθηκαν στην Αυστρία και ίσως για το ένα το θυμάστε η πολιτιστική πρωτεύουσα του 2009 στο Λίντς. Χάρη στην τοπική αυτοδιοίκηση και η πόλη και η περιφέρεια από πολλών ετών είχε στραφεί προς ευρωπαϊκά θέματα και όταν ε, καθορίστηκε πολιτιστική πρωτεύουσα ε, με τον τίτλο ε, «Το αλλαγμένο Λίντς» μεταμορφώθηκε σε μία σύγχρονη πολιτιστική πρωτεύουσα. Ο πολιτισμός και ο τουρισμός και αυτό το θέμα μπόρεσε να προωθηθεί σε τέλεια συμβίωση κατά αυτή τη διάρκεια και τρία χρόνια τώρα μετά την πολιτιστική πρωτεύουσα βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμη μία δυναμική και μία ανάπτυξη στο χώρο αυτό. Επίσης όσον αφορά τον τουρισμό ε, είχαμε ε, ε, πρωτοβουλίες στο χώρο Φοράντλμπερκ την ορεινή αυτή περιοχή όπου ε, είχαν δημιουργηθεί διάφορες δραστηριότητες ε, πληροφόρηση για εκδηλώσεις ε, τρόπο οργανώσεως εκδηλώσεων και διάφορες άλλες πολιτιστικές πρωτοβουλίες και όσον αφορά την συγχρηματοδότηση βλέπουμε ότι και η πρωτεύουσα της Αυστρίας η Βιέννη έχει συμβολή στην κατάρτιση του δικτύου από το Μπέλφαστ, το Μπιλμπάο μέχρι τη Σόφια μέσω Βιέννης κατά ώστε να υπάρχει μία άμυλα μεταξύ των διαφόρων περιοχών και ε, βλέπουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο ε, ο πολιτισμός και η δημιουργική κλάδη μπορούν να συμβάλλουν στην έπτυξη ανάπτυξη ε, με εξυπνάδα στην Ευρώπη και χωρίς εντάσεις. Και ακριβώς στην σημερινή εποχή όπου οι δημόσιοι πόροι είναι περιορισμένοι και οι οικονομικές συνθήκες δύσκολες θα πρέπει να μπορέσουμε να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες όλων των τομέων δηλαδή και η τέχνη και, ο πολιτισμός πρέπει να εδρεωθούν στη στρατηγική της Ευρώπης και το ίδιο ισχύει και για τα λειτουργικά προγράμματα των μεμονωμένων ε, χωρών ε, σε εθνικό επίπεδο. Κυρίες και κύριοι, ε, είμαι, έχω πλήρη συνείδηση ότι εδώ υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και ιδίως να πείσουμε τους πολιτικούς. Αλλά πιστεύω ότι από κοινού θα το καταφέρουμε. Και προς εσάς κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ε, θα μπορέσετε ε, να συμβάλλετε και εγώ σαν υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο και να σας πω ποια είναι τα βασικά προγράμματα για, ε, που έχουν προτεραιότητα για τον άμεσα επόμενο χρόνο κατά τρόπον ώστε να διαργανώσουμε κοινέ δραστηριότητες με την περιφέρεια. Υπάρχουν ορισμένα προγράμματα που έχουν ήδη ε, καταρτιστεί για την ε, Αυστρία, την ψηφιοποίηση των περιφερειακών ε, σινεμά και στον τομέα της επαγγελματικής αντιμετώπισης του δημιουργικού τομέα στο σύνολό του μία θερμή επιθυμία και ευχή προς εσάς κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές είναι να μπορέσει να υπάρξει καλύτερη προβολή του πολιτισμού και της τέχνης στην Ευρώπη και από κοινού να συμβάλλουμε ώστε και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ο πολιτισμός να αποτελέσει ένα παράγοντα ανταγωνιστικότητος και συνοχής διότι ο Ζακ Ντολόρ είχε πει ότι κανείς δεν ερωτεύεται μία κοινή αγορά. Αυτό που προσπαθούσα να πει είναι ότι ο πολιτισμός είναι μία παράβατη αξία και θα πρέπει σε όλους τους πολιτικούς τομές, τομείς να χρησιμοποιούμε αυτή τη δύναμη ε, της τέχνης και του πολιτισμού και σας ευχαριστώ. Thank you, Madam Ελπίζω να δεχτείτε μερικές ερωτήσεις ή σχόλια από τους βουλευτές. Η Κωνσταντσα Κρέλ. Πρώτη. άλλωστε εκείνη ήταν η εμπνεύστρια της ιδέας να καλέσουμε την κυρία Υπουργό, πρώτα η Κωνσταντσα και μετά η άλλη. Ε, λέει ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ Χαίρομαι πάρα πολύ που τα καταφέρατε και ήρθατε. Δεν παραβιάζετε παρανοιχτές θύρες ε, εμένα σε ότι ε, είπατε ότι θα πρέπει να προωθηθεί ο πολιτισμός. Ξέρω πολλά πολιτιστικά σχέδια, ιδιαίτερα στα κρατήδια Μπούργκελαντ και στη Σαξονία. Και στο Μπούργκελαντ είναι και διασυνοριακό το πρόγραμμα αυτό Αυστρίας-Γερμανίας και συνεργαζόμαστε καλά. Το γεγονός ότι είστε Ομοσπονδιακή υπουργό με κάνει να σας ρωτώ το εξή. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ συχνά μας κοπανάνε συνέχεια την περίφημη λέξη επικουρικότητα. Ιδιαίτερα όταν βολεύει αυτόν που τη χρησιμοποιεί κάθε φορά. Ξέρω λοιπόν ότι για τον πολιτισμό είναι πάρα πολύ της μόδας και αγαπούν πολύ αυτή την έκφραση οι ενδιαφερόμενοι. Βέβαια, όχι όταν πρόκειται να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πολιτιστικά. Λοιπόν, στο Συμβούλιο εσείς Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς επιχειρηματολογείτε ότι ο πολιτισμός δεν είναι απλώς υπόθεση της επικουρικότητας των κρατών μελών, αλλά είναι και ευρωπαϊκό ε, ζήτημα. Εγώ διέτρεξα λίγο τη σύνοψη της μελέτης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πιο συγκεκριμένα έχετε να μας πείτε κάτι για το δημιουργικό τομέα και πώς επηρεάζει την αγορά εργασίας γιατί για μας θα μας βοηθούσαν τα επιχειρήματα γιατί είναι και κοινωνικό το όφελος ας πούμε και από τα διαρθωτικά ταμεία για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ευχαριστώ. Ο Γιάνν Όλμπριχτ. Ευχαριστώ. Υπουργέ, για την παρουσίαση αυτή, για την εμπειρία σας που μοιραστήκατε μαζί μας. Έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Εγώ είμαι συγγητής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με πιέζουν εδώ και μήνες ε, οι δημιουργοί, οι καλλιτέχνες, να βάλω κάτι στον κανονισμό. Αν δείτε τον κανονισμό δεν γίνεται ιδιαίτερος λόγος για τον πολιτισμό ε, στο Περιφερειακό Ταμείο. Τι θα προτείνει η Αυστρία λοιπόν στο Συμβούλιο, γιατί μέχρι τώρα είναι πολλά τα στοιχεία. Πρώτον, μπορούμε να εισαγάγουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες καλλιτεχνικές ε, δραστηριότητες. Αλλά κάπου να το λέει αυτό, γιατί για να αποκλείεται δεν μπορεί. Υπάρχει το άρθρο 3, το πεδίο στήριξης, είναι επενδύσεις στην παιδεία, στην υγεία και στα κοινωνικά. Τα κοινωνικά ε, εμπεριέχουν τον πολιτισμό ή όχι. Αλλιώς, πού θα το βάλουμε, αν δεν τον περιέχουν τον αποκλείουν και στις επενδυτικές προτεραιότητες ένα είναι το σημείο που αναφέρει την πολιτιστική κληρονομιά και τίποτα άλλο, τελεία. Δηλαδή, α, και κατά τα άλλα, συμμερίζομαι την άποψή σας ότι η επένδυση στον πολιτισμό το 2020 είναι ε, κομβική σημασίας, γιατί επενδύουμε στα μυαλά των νέων γενεών κτλ. Ωραία. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά πού θα προτείνετε στο Συμβούλιο να μπει συγκεκριμένα στον κανονισμό για να συνεργαστώ μαζί σας. Προς το παρόν δεν μου είναι τόσο εύκολο, γιατί δεν ξέρω τα συγκεκριμένα. Σηκώστε τα χέρια σας, γιατί δεν έχουμε σημειώσει όλα τα ονόματα. Γιάννης Νίλσεν. Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας και για τα όσα μας είπατε. Έχω την άποψη ότι έχετε δίκιο, είστε στο σωστό δρόμο και ο πολιτισμός είναι σημαντικός. 15 χρόνια είμαι δήμαρχος και ξέρω ότι όταν δεν συμπεριλαμβάνεται ο πολιτισμός δεν μπορεί να πετύχει καμία προσπάθεια στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, γιατί είναι τμήμα αυτού. Αλλά η δομή της διαρθωτικής πολιτικής είναι ευρωπαϊκές αξίες ο στόχος και από εκεί και πέρα, από κάτω προς τα πάνω, χρειάζεται να πείσετε σε κάθε περιφέρεια για το τι είναι το πιο σημαντικό να γίνει. Την Παρασκευή. Συναντήθηκα με τον Έμιλο, ο οποίος ε, θα είναι ε, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής ε, Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2013 και ε, που βεβαίω θα θελήσει να προωθήσει και όλα τα πολιτιστικά θέματα. Και στη δικιά μας ε, περιοχή είπαμε ότι και ο αθλητισμός είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θα πρέπει να ε, συμμετάσχει σε αυτή την πολιτιστική διαδικασία που τελικά θα δημιουργήσει θέσεις εργασία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βεβαίω ο πολιτισμό μαζί με όλα τα άλλα σημαντικά ζητήματα θα πρέπει να έχει σημαντική θέση. Ο κύριο Στάγκλερ παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν ε, κυρία ε, Υπουργέ, θέλω να σας συγχαρώ για την ε, έκθεση αυτή καθώς και του συντάκτες της διότι είναι μια καλή βάση επί της οποίας μπορούμε να συζητήσουμε για την δημιουργική οικονομία και για την περιφερειακή ανάπτυξη. Βλέπουμε βάση των αριθμών που για τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αυστρία ότι μπορεί κανείς να επηρεάσει την περιφέρεια αν γίνει η προσπάθεια διότι βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό ε, ένα μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που είχε προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήταν 1,7 χρησιμοποιήθηκε ή στην περιφέρεια της Αυστρίας με πολύ καλό αποτέλεσμα και βλέπουμε ότι ουσιαστικά το Ταμείο ΕΦΡΑ είναι αυτό το, δηλαδή ε, το, Περιφερειακό Ταμείο είναι αυτό το οποίο συμβάλλει και είναι σημαντικό και αυτό ήταν έκπληξη για μένα γιατί ε, νόμιζα ότι υπήρχε μία ε, εμπλοκή της γεωργίας στην περιφερειακή στη περιφερειακή πολιτική. Ε, αλλά είδαμε ότι το περιφερειακό ταμείο για, τον, ε, για την ανάπτυξη ε, δεν έδωσε τη δέουσα σημασία και υπάρχουν ακόμη πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες. Ως αυτό που είπε ο Γιάννα Άλμπριχτ έχω να το υπερθεματίσω διότι πιστεύω ότι στο μέλλον θα πρέπει να δούμε πώς θα ρυθμίσουμε το θέμα των ταμείων διότι από πλευράς τέχνης βλέπουμε ότι υπάρχει πολλές φορές μία έμεση εμπλοκή η οποία δεν αντιμετωπίζεται ε, ευθέως και θα μπορούσαμε να έχουμε στηρίξει καλύτερα στον τομέα της τεχνολογίας στην περιφέρεια ε, και όσον αφορά και την ε, ε, ανανέωση, την ανάπτυξη. Εάν θέλουμε λοιπόν όντως να προχωρήσει η ανάπτυξη πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις περιφερειακές δράσεις σαν προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και όσον αφορά την κινητικότητα θα πρέπει επίσης να θεωρήσουμε ότι υπάρχει περιφερειακά μία διασυνοριακή συνεργασία και όσον αφορά τις επενδύσεις και την παιδεία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πόρους από το Ταμείο Συνοχής και πρέπει να δούμε ε, βάσει αυτής της εκθέσεως και των προτάσεών της πώς μπορεί κανείς ε, να βελτιώσει την, ε, το στρατηγικό προγραμματισμό. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ο πρώτος στόχος, δηλαδή να υπάρχει μία προώθηση της περιφερειακής πολιτικής. Είναι κάτι που πρέπει να απαχοσχολήσει εμάς. Επίσης, ε, όσον αφορά αυτό που κάνουν μόνες τους οι χώρες, πιστεύω Κύριε συνάδελφε, δεν μπορούμε να, να συνεχίσουμε τόσο πολύ. Τελευταία φράση. Ε, η συνεργασία είναι ένα θέμα των χωρών, αλλά θα μπορούσε να συντονιστεί καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε άλλους τέσσερις που θέλουν να ρωτήσουν. Σας παρακαλώ, όσο γίνεται πιο σύντομο. Η Μαρίτε Σάντσης και μετά ο κύριος Χρυσόγελος. Δύο-τρεις πληροφορίες ήθελα να δώσω. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Κράνης που ε, ε, πρότεινε στην, και προσκάλεσε την κυρία Υπουργό. Έχουμε κάποια στοιχεία. Το 2008 παρουσίαζαν 860 δισεκατομμύρια τζίρο και 14 εκατομμύρια 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Ε, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό κλάδο. Πρέπει οπωσδήποτε να διευρυνθεί η λεγόμενη βιομηχανία της δημιουργίας. Ε, κυρίως βάσει του σημείου 6. Ε, εγώ ζω και προέρχομαι από τα γαλλο-ισπανικά ε, σύνορα. Έχουμε λοιπόν επενδύσει 32 εκατομμύρια ευρώ σε ένα θέατρο διασυνοριακό το οποίο αποτελεί ε, ένα πάρα πολύ ζωντανό πυρήνα σκέψης, ανταλλαγής και τα λοιπά θεατρικέ Κάνει, θεατρικές παραστάσεις στο θέατρο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να ε, πιέσετε κι εσείς έτσι ώστε να ληφθεί περαιτέρω και περισσότερο οπωσδήποτε υπόψη το θέμα του πολιτισμού. Ε, ο κύριος Χρυσόγελος. Είμαι πεπισμένο ότι τα θέματα του πολιτισμού και της τέχνης είναι πάρα πολύ σημαντικά, όχι μόνο για την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και για την κοινωνική συνοχή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή: Αν έχετε ετοιμάσει κάποιες συγκεκριμένες όμως προτάσεις για το Ταμείο Συνοχής, για πολιτιστικά ζητήματα, Μα δεν είναι θέμα της Αυστρίας, ευτυχώς, λέει η Πρόεδρος, ο κύριος Τσέλε. Ευχαριστώ κυρία Ομοσπονδιακή Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Ακριβώς δείχνουν τα όσα κάναμε μέχρι τώρα στο Βερολίνο, δηλαδή ενίσχυση και προώθηση ιδιαίτερα της δημιουργικής ε, ε, δραστηριότητας και του πολιτισμού με ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν μιλούμε για ε, κρατικά θέατρα ή όπερες, τα κτίρια, αλλά ενίσχυση των δημιουργών ε, σε μια τέτοια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για να μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό στο Βερολίνο το συνδέσαμε ως εξή. Έχουμε την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη και χρειάζεται ευελιξία στα κονδύλια και τα ταμεία. Έχει προκύψει μεγάλη βιομηχανική έρημος γιατί έχουν φύγει τα εργοστάσια και είναι εργατικές κατοικίες, ε, συνοικίες ολόκληρες. Εκεί χρειάζεται σήμερα ανάπλαση. Ε, και από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Κοινωνικό Ταμείο για την απασχόληση και ε, έτσι οδηγήθηκαν σε αυτές τις περιοχές οι καλλιτέχνες και οι περιοχές αναβαθμίστηκαν άρδιν. Πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες έγιναν δύο ή τρία χρόνια μετά την αρχική ε, χρηματοδότηση και μετά αυτή την πρώτη μαγιά που τους δώσαμε κατέφεραν ε, να αναπτυχθούν μόνοι τους και να αυτοχρηματοδοτούνται. Αυτό είναι ο στόχος της ε, πολιτικής και δεν έχω ερώτηση αλλά παράκληση. Εσείς μπορείτε να μεσολαβήσετε στην κυβέρνησή σας να μας υποστηρίξει να υπάρχει ευελιξία προσαρμογή των ταμείων στις περιφερειακές ανάγκες και για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Στο Βερολίνο έχουν αποφεληθεί και εργάζονται εκεί 100.000 άνθρωποι. Είναι μεγάλο το δυναμικό και ο παλμός και η ελκυστικότητα της πόλης. Ο κύριος Αλφονζή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα για να ευχαριστήσω βεβαίως την κυρία Υπουργό ε, Σμιτ ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό της πολιτιστικής δραστηριότητας ως οχήματος ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε εν μέρη υπόψη το σημείο αυτό, αλλά δεν είναι αρκετό. Ε, έχει ασχοληθεί περισσότερο με το κατά κάποιο τρόπο νεκρό πολιτιστικό ε, κεφάλαιο, ενώ υπάρχει ένα πολύ ζωντανό και ζών ε, κεφάλαιο, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, μας απασχολήσει. Βεβαίως είναι πιο εύκολο να χρηματοδοτήσει κανείς την οικοδόμηση ας πούμε ενός πολιτιστικού, ε, ε, μιας πολιτιστικής υποδομής ε, παρά αυτή την άειλη υποδομή. θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Τέλος, το ενδιαφέρον της χρήσης του Ταμείου Συνοχής για τέτοια πολιτιστικά στοιχεία είναι σημαντικό ε, το ότι θα πρέπει να γίνουν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο κυρίως και ότι θα πρέπει να φύγει από την κεντρική κυβέρνηση ε, αυτού του είδους ε, η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάντσμα. Δεν σας είχα δει προηγουμένω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ποριέ. Νομίζω ότι είστε σε μια πολύ κρίσιμη και σημαντική φάση των συζητήσεων στην Επιτροπή μας, γιατί αυτό που χρειάζομαστε πάντα είναι αριθμοί, στοιχεία, γεγονότα. Και ακριβώς ο πολιτισμός και ο δημιουργικός κλάδος συχνά θεωρείται κάτι που απλώς κοστίζει δαπανηρό, ενώ σήμερα μας δώσατε μια σειρά αποδείξεων ότι αποφέρει και κέρδος και νομίζω ότι ε, αυτό είναι υπέρ των διαφθορτικών μας ταμείων. Αυτό που θέλουμε βεβαίως είναι πρώτα συνοχή και κοινωνική ένταξη, αλλά τα δικά σας παραδείγματα έδειξαν ότι ε, πιάνουν τόπο τα χρήματα και για εκείνους που ασχολούνται με τα θέματα της δημιουργίας και του πολιτισμού και στο μέλλον σας παρακαλώ να ε, συνεχίζετε να συνεργάζεστε με τον Επίτροπό μας κύριο Χάν και με τον ε, Επίτροπο για τη Γεωργία, έτσι ώστε οι ιδέες αυτές να μην πάνε χαμένες, αλλά να συμπεριληφθούν και ε, στις δικές τους προτάσεις με σθένος και ρητά. Ευχαριστώ πολύ. Υπουργός, να απαντήσω στα διάφορα θέματα. Τη συζήτηση για την επικουρικότητα βεβαίω τη γνωρίζουμε και στο εσωτερικό της Αυστρίας. Έχετε απολύτω δίκιο. Κυριαρχεί πάντα στη συζήτηση και στις απόψεις του καθενός. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθούμε στα διάφορα έργα να περιγράφουμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Παράδειγμα, διεθνή συνεργασία ή Κάτι άλλο που κάνουμε και σε άλλους τομείς πολιτικής στην οικονομία, το συνδέουμε με την απασχόληση και με την οικονομική δυναμική. Αυτό είναι το επιχείρημα. Το είπατε κι εσείς. Ε, μιλήσατε για ένα μετασχηματισμό και ανάπλαση παλιών βιομηχανικών εγκατελειμμένων περιοχών. Ακριβώς αυτό έγινε στο Λίντς 30.000 θέσεις απασχόλησης δημιουργήθηκαν σε παλιές ενοικίες και γειτονιές υποβαθμισμένες εντός εισαγωγικών. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυναμική για ένα μετασχηματισμό, ε, μεταμόρφωση ουσιαστική των πόλεων και της οικονομίας. Οπότε αυτό δεν θα το έφερνα το ένα αντιμέτωπο με το άλλο. Συνδυάζονται αυτά πάρα πολύ και με μεγάλη αυτοπεποίθηση όχι, και ε, ο πολιτισμός και η τέχνη έχουν και οικονομικά, όχι μόνο, αλλά και οικονομικά επιχειρήματα. Γιατί καμιά φορά αυτό δεν αναδεικνύεται στη συζήτηση. Διστάζουμε. Εγώ λέω ότι δεν το χρειάζεται πολλές φορές ο πολιτισμός και η τέχνη γιατί είναι τόσο δυναμικοί κλάδοι και δημιουργούν τόσες απασχόλησεις που δεν χρειάζεται αυτό το επιχείρημα. Ε, αναφερθήκατε στην τέχνη και τον πολιτισμό ως ε, ένα θέμα εγκάρσιο, δηλαδή που εντάσσεται σε όλους τους τομείς πολιτικής. Αλλά δεν μου αρκεί αυτό, συμφωνώ με τον κύριο Στάτλερ. Θα πρέπει αυτός ο δημιουργικός τομέας να γίνει πιο ορατός, να του δώσουμε μεγαλύτερη προβολή και στους κανονισμούς μας και στον κανονισμό για το Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης. Εγώ δεν έχω αυτή τη στιγμή ολοκληρωμένη πρόταση, αλλά κατά την άποψή μου οι υποδομές πολιτισμού θα πρέπει να συμπεριληφθούν βεβαίως όπως και η πολιτιστική προσφορά. Αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να τα προωθήσουμε, να τα φέρουμε στο προσκήνιο και να μην λέμε ότι είναι ένα θέμα που αφορά ε, όλες ε, τις πολιτικές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μικρομεσαίες είναι αυτές οι επιχειρήσεις, έτσι κι αλλιώς. Ε, δεν πειράζει να το έχουμε αναφέρει δύο φορές. Καλύτερα δύο φορές παρά να το αποσιωπούμε. Και αυτόν τον τομέα, την τέχνη, τον πολιτισμό, τη δημιουργία. Θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να εργαζόμαστε ταυτόχρονα σε διάφορα επίπεδα και στο εθνικό επίπεδο, η διαδικασία της ανάπτυξης στρατηγικής, δηλαδή των στρατηγικών προγραμμάτων των κρατών μελών, αλλά θα πρέπει ήδη να προγραμματίζουμε και να προετοιμάζουμε και το περιφερειακό επίπεδο. Γιατί εκεί στις ομάδες εργασίας μπαίνουν τα θεμέλια για αυτά και από εκεί και πέρα βέβαια το μεγάλο επίπεδο το νομοθετικό πάνω από τα άλλα δύο. Και εδώ πραγματικά ποντάρω ειλικρινά σε εσά και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπουν τα θέματα αυτά στη νομοθεσία. Η πρωτοβουλία, ε, η δέσμευση, η στράτευση έτσι κι αλλιώς θα έρθει από την περιφέρεια, από τους ίδιους τους ανθρώπους. Αλλά χρειάζονται την αναγνώριση, την ένταξη και την ενσωμάτωσή τους και στα τεχνικά ζητήματα, στη νομοθεσία, ας πούμε, στον κανονισμό για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και γι' αυτό θα φροντίσω, θα ασχοληθώ και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίδετε να το συζητήσω μαζί σας. Ε, και για μένα είναι ιδιαίτερη εμπειρία αυτή. Σας ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως εμείς σας, θα σας στηρίξουμε, αλλά θέλουμε να δουλέψετε και με το Συμβούλιο και με την ε, Κομισιόν έτσι ώστε να βοηθήσουμε την Ευρώπη που χρειάζεται πλέον νέα ε, οχήματα που θα την οδηγήσουν προς την ανάπτυξη, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας κτλ. Θα πρέπει να δούμε πώς είναι δυνατόν να σταχυολογήσουμε στα πλαίσια της πολιτιστικής ανάπτυξης ε, αυτά τα δυναμικά στοιχεία τα οποία μπορούν να δώσουν μια νέα όθηση και στην οικονομία, δημιουργία θέσεων εργασία κτλ. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την έμπνευση που μας δίνετε. Σίγουρα μας ανοίξατε την όρεξη, λέει η Πρόεδρος, για να συνεργαστούμε, να δουλέψουμε μαζί με την Αυστρία. Ευχαριστούμε πολύ.